So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα μπορούν να το κάνουν. Hey Nacho, can you go outside? I'm not starting the meeting until δεν θα, δεν αρχίσω αυτή τη συνεδρίαση μέχρι να καθίσετε όλοι. Όλοι οι συνάδελφοι, κυρία Λαλού. Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Καλώς όρισμα θερμά τον κύριο Σικλούνα, που είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σας προσκαλέσαμε γιατί θα θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψεις για την στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Συρία και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τη διαδικασία της Γενέβης και να, επαρκές, ε, να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο για την αποδοχή της δημοκρατικής διαδικασίας. Δύο παρατηρήσεις. Κάποια ε, αραβικά κράτη έχουν ξανανοίξει τις ε, πρεσβείες του στη Δαμασκό και προσπαθούν να εξομαλύνουν τις διπλωματικές σχέσεις με πλήρη αναγνώριση. Ο Αραβικός Σύνδεσμος μπορεί να δεχθεί τη Συρία στα μέλη του ξανά και επίσης ο ΙΕ ε, προσπαθεί να στηρίξει την διαδικασία της Γενέβης, ενώ υπάρχει ε, μεγάλη απογοήτευση από πολλούς και από εμά για αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ επισφαλής η θέση στη Συρία και όλο και περισσότερες ε, πολιτοφυλακές με την ε, υποστήριξη του Ιράν μπαίνουν στην Συρία. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συρία αυτή η τρίτη διάσκεψη για τη Συρία ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ε, την κοινωνία των πολιτών ε, και στην Τουρκία και να τους δώσει τα επαρκή εργαλεία και επίσης τι μπορούμε να περιμένουμε από τη στάση του Αραβικού Συνδέσμου απέναντι στη Συρία. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις από πλευράς μου. Οι συνάδελφοι θα έχουν πολλές ακόμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις με την Επιτροπή σας. Έχουμε καθυστερήσει. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο να τον πιο σύντομος, παρότι το θέμα της Συρίας ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα σε τρία τμήματα. Καταρχάς, να σε ενημερώσω για την κατάσταση επιτόπου. Δεύτερον, να δούμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θέσεις ε, της ε, διεθνούς κοινότητας και τέτοιο. Και τρίτον, την προετοιμασία τι μπορούμε να κάνουμε για την προετοιμασία της τρίτη διάσκεψης τη Βρυξέλλας για τη Συρία. Η κατάσταση στη Συρία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση εντό τη Συρίας ε, ως ε, επιστροφή στην ομαλότητα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν λιγότερες μάχες ε, στη Συρία από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η κατάσταση στη Συρία δεν μπορεί να θεωρηθεί, δεν μπορεί να περιγραφεί και να θεωρηθεί ομαλή. Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις που είχαν σημασία μεγάλη ήταν η αναγγελία από τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν τα στρατεύματά τους από την βορειοανατολική Συρία. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα σε ποιο βαθμό και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί η αποχώρηση, όμως οι επιπτώσεις απόφασης αυτής ε, γίνονται αισθητές ε, στη Συρία. Καταρχάς, οι κουρδικές δυνάμεις οι οποίες ε, υποστηρίζονταν τις ΗΠΑ βρέθηκαν σε μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να επενεκτιμήσουν τη θέση τους και ένα από τα μέτρα τα οποία έλαβαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση είναι να έρθουν ξανά σε επαφή με το καθεστώς ε, που μέχρι τότε ήταν ορκισμένοι εχθροί του. Επίσης, οι ακραίες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, ειδικά ο ISIS, ε, και παρότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι θα επιστρέψουμε στην κατάσταση όπου το Ισλαμικό λεγόμενο κράτος που κάλυπτε, θα καλύπτει πάλι τμήματα της Συρίας, όμως ε, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ακραίες ομάδες, οι εξτρεμιστικές ομάδες είναι όλο και πιο δυνατές και ανακτούν θέσεις ε, στο εσωτερικό της χώρας. Φυσικά, μια άλλη οντότητα που ενισχύθηκε την απόφαση των Αμερικανών είναι το καθεστώς, γιατί τώρα είναι σε μια θέση όπου οι αντίπαλοι τους, οι Κούρδοι ας πούμε, χρειάστηκε να αλλάξουν θέση και να έρθουν σε επαφή μαζί τους η παρουσία των Αμερικανών, Αμερικανικών στρατευμάτων που σήμαινε τη δυνατότητα άμεσης ε, αντίδρασης, δεν θα υπάρχουν πια αυτές οι δυνάμεις, ε, βραχυπρόθεσμο, και αυτό ενίσχυσε τη θέση του καθεστώτος και των υποστηρικτών, κυρίως ε, της Ρωσίας και του Ιράν. Όπως είπα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα λάβει η χώρα αυτή η αποχώρηση των δυνάμεων. Ε, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα. Θα γίνει μια συνάντηση της Συμμαχίας για την Αντιμετώπιση στο, του ISIS στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Ε, συμμετέχουμε σε αυτή τη συμμαχία. Συνεργαζόμαστε πάνω σε μια σειρά μέτρων, ενός πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστούν στην ε, επόμενη συνεδρίαση της συμμαχίας. Φυσικά, η υλοποίηση αυτών των μέτρων ε, εξαρτάται από την ικανότητά μας να βρούμε εταίρους, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη Συρία, ε, που θα, κάλυπταν, που θα μας κάλυπταν και θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν τώρα όμως κάποιες αμφιβολίες για το πόσο μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν λιγότερες μάχες, το είπα. Όμως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία είναι πολύ ευπαθής, πολύ ευάλωτη, όπως και πριν. Ε, καταφέραμε να αποτρέψουμε μία φοβερή καταστροφή στο Ιντλίμπ. Εν μέρη χάρη στην συνεννόηση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να αισθανθούν ότι έκαναν κάτι ε, για αυτή τη διαμεσολάβηση Τουρκίας και Συρίας για να θα καταφέρουν να συνοηθούν και ενώ αποτρέψαμε την ανθρωπιστική κρίση, ο κίνδυνος επιδείνωσης κατάστασης δεν έχει φύγει. Αναφέρατε, Πρόεδρε, την τάση εξομάλυνσης με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Ισχύει αυτό. Κάποιες ε, αραβικές χώρες έχουν ξανανοίξει τις πρεσβείες τους στη Δαμασκό, κάποιες ε, αερογραμμές, αεροπορικές, αεροπορικές εταιρείε ε, πετάνε ξανά στην Δαμασκό, συνεδριάσεις γίνονται. Την περασμένη εβδομάδα ένα οικονομικό φόρουμ έγινε στο Ντουμπάι ε, για την ε, Συρία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει βαθμιαία εξομάλυνση των σχέσεων. Ξεκαθαρίσαμε και εδώ συμφωνούμε με τις ΗΠΑ ότι είναι μια εξομάλυνση που πιστεύουμε ότι είναι άκερη. Καταρχάς, γιατί το καθεστώς δεν έκανε τίποτα για να αξίζει αυτή την αναγνώριση, δεν έκανε καμία παραχώρηση, δεν έχει έρθει σε επαφή με τη διεθνή κοινότητα με οδήποτε τρόπο, δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι επιθυμεί να έχει σχέσεις. Επομένως, η εξομάλυνση θα ήταν ένα βραβείο σε ανταλλαγή, για αντάλλαγμα ποιου πράγματος που έδωσε το καθεστώς. Τίποτα του τίποτα. Θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αυτό το μήνυμα, μόνο που τελικά τα αραβικά κράτη θα αποφασίσουν και θα καθορίσουν τι σχέσεις θέλουν να έχουν με τη Συρία. Και κυρίως αυτές θα αποφασίσουν αν επιθυμούν να ξαναφέρουν τη Συρία στον Αραβικό Σύνδεσμο. Ετοιμάζουμε και μια Υπουργική Σύνοδο με, την, με τα κράτη ε, του Αραβικού Συνδέσμου στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα και μια συνοκορυφής που θα γίνει στην Αίγυπτο ε, τέλη Φεβρουαρίου και φυσικά αυτό είναι από τα βασικά θέματα που στέλνουμε και ε, μηνύματα που στέλνουμε στους Άραβες εταίρους. Αυτή την ευρωπαϊκή θέση παρά τις πολλές προκλήσεις, παρά τις εκδηλώσεις και τα γεγονότα επιτόπου και αλλού, αυτή η ευρωπαϊκή θέση είναι απαρασάλευτη και βασίζεται όχι μόνο σε αρχές, αλλά και σε σωστές πολιτικές απόψεις και στεναρές πολιτικές απόψεις. Από τη μία λοιπόν, δεν πρέπει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις σε αυτή τη φάση, να μην κάνουμε ανοικοδόμηση μέχρι να υπάρχει μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία στη Γενέβη με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τρίτο, το θέμα των επιστροφών των προσφύγων το οποίο είναι ένα επίμαχο θέμα, γιατί φυσικά πολλοί από εμά ε, συμφωνούμε ότι θα θέλαμε οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στις αιστείες τους, οι ίδιοι οι πρόσφυγες το επιθυμούν, όμως ε, αυτή η επιστροφή θα πρέπει να λάβει χώρα ε, στο σωστό πλαίσιο, δηλαδή να είναι ασφαλής, αξιοπρεπής και επιθυμητή. Υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές στο ΙΕ που ξεκαθαρίζουν πώς οι επιστροφές λαμβάνουν χώρα και όταν ακούμε από διάφορους φορείς ότι οι συνθήκες είναι όριμες και σωστές να αρχίσουν να επιστρέφουν οι πρόσφυγες, η δική μας απάντηση πάντα ήταν αποδείξτε το. Δείξτε μας ότι υπάρχουν σωστές συνθήκες, ούτως ώστε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Γιατί όταν βλέπουμε την κατάσταση στη Συρία, βλέπουμε ότι το καθεστώς υιοθετεί κάποια κάποιους νόμους για να στερήσει τις περιουσίες από τους πρόσφυγες. Η κατάσταση ασφάλειας είναι τέτοια όπου δέχονται εκφοβισμούς και διακρίσεις όσοι επέστρεψαν στις αιστείες τους και επομένως όλα αυτά μαζί μας δείχνουν και δεν μας πείθουν ότι συντρέχουν οι συνθήκες για την επιστροφή τους. Συνεχίζουμε λοιπόν να θεωρούμε ότι η θέση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Απριλίου του 2018 εξακολουθεί να ισχύει. Είχαμε θέση ε, απόψη, ανταλλαγής απόψεων με τα κράτη-μέλη για, την, ε, για αυτές τις απόψεις. Στην άτυπη Υπουργική Υπουργών Εξωτερικών συζητήσαμε το θέμα και δεν βλέπουμε ότι υπάρχει λόγος να αλλάξουμε αυτή τη θέση ε, προς το παρόν. Τέλος, δύο λόγια για την ε, τρίτη διάσκεψη των Βρυξελών, όπου αποφασίσαμε ξανά ότι έχει νόημα να γίνει αυτή η διάσκεψη, να καλέσουμε λίγο πολύ τους ίδιους ανθρώπους με το παρελθόν, να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στο πολιτικό επίπεδο, ε, ένα πλαίσιο δηλαδή για τη διαδικασία του ΟΗΕ, να εστιάσουμε στα ανθρωπιστικά και στη δέσμευση ε, να δώσουμε βοήθεια στους πρόσφυγες της, της ε, του Σύρους εντός της ε, Συρίας και στις ε, γειτονικέ χώρες και να βοηθήσουμε τις γειτονικέ χώρες. Έμφαση στην κοινωνία των πολιτών θα είναι μια ημέρα διαλόγου. Η... Θα υπάρχει και υπουργική σύνοδος για το ρόλο της ε, κοινωνία των πολιτών και το ρόλο των γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σικλούνα αυτές τις ε, αρχικές σας παρατηρήσεις. Τώρα θα συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων. Έχουν ζητήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι. Κύριε Σπανιό, κύριε Λόχπιλερ και ε, ε, κύριε... Έχω ξεχάσει, κύριε Βαλόντ, και ο πρόεδρος επίσης. Πέντε ομιλητές λοιπόν, 1,5 λεπτό ο καθένας. Σας ξεκινήσουμε με τον κύριο Παγνιό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Αναπληρωτή, Τελεξική Διευθυντή, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η παρουσίαση που κάνατε μας δείχνει ότι η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη και στρατιωτικά και πολιτικά και ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση σε κανένα από τα δύο επίπεδα συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτό φάνηκε από αυτά που είπατε, όμω ε, δεν αναφερθήκατε σε κάτι κατά την άποψή μου. Σημαντικό είναι η κατάσταση των Κούρδων στην Συρία. Η προστασία του πληθυσμού του Κουρδικού είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε ότι ήταν από του σημαντικότερου συμμάχου μα στη μάχη κατά του ΆΙΣ. Και φαίνεται ότι του έχουμε παραμελήσει μετά από την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων και με την πολιτική της Τουρκίας. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή κινδύνους να ε, τους απειλούν. Φαίνεται ότι η προτίμηση ε, των Τούρκων θα ήταν να δημιουργηθεί ένα προτεκτοράτο αρχικά και τελικά τα στρατεύματά τους να αναπτυχθούν στην περιοχή την κουρδική της Συρίας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να μας ανησυχήσει το ζήτημα αυτό, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των Κούρδων στη Συρία. Η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει από τον πρόεδρο Ερδογάν να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των Κούρδων, αλλά τώρα αναρωτιέται κανείς, μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη του κυρίου Ερντογάν. Περνάμε λοιπόν από μια στρατιωτική περίοδο σε μια περίοδο πολιτικών ε, λύσεων και εξελίξεων και σε αυτήν την νέα περίοδο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της ασφάλειας των Κούρδων. Ευχαριστούμε κύριε Ανταλόν. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο Ιντλίπ πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των πιο πλέον εξτρεμιστικών ομάδων και θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ότι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον στην πόλη αυτή. Και δεύτερον, πιστεύω ότι θα είχε μια κάποια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επαφή με το καθεστώς Ασάντ, αν μη τι άλλο για να φροντίσουμε να μην απελευθερωθούν όλοι εκείνοι οι τζιχαντιστές που βρίσκονται σε κουρδικές φυλακές, φυλακές του κουρδικής περιοχής και να απελευθερωθούν και αυτοί να γνωρίζουμε πόσες χιλιάδες είναι, αρχίσουν να κυκλοφορούν. Αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο κίνδυνο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων στο μέλλον και προ ενός μεγάλου κινδύνου. Σας ευχαριστούμε κύριε Λοχπίλαρ. Τρεις ερωτήσεις. Στην τελευταία διάσκεψη των δωρητών έγιναν δεσμεύσεις για 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται δεσμεύσεις ανάλογες και φέτος. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι αυτό το οποίο υπογραμμίστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σαφή θέση ότι θα δοθεί βοήθεια για νοικοδόμηση στην Συρία όταν υπάρξει μια συνολική πολιτική μετάβαση. Αλλά τώρα στην δουλειά που γίνεται ήδη επί τόπου. Μπορεί να γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και των σχετικών υποδομών και ανοικοδόμησης και τέλος λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να έρθουν οι εγκληματίες πολέμου ενώπιον της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ. Τις προάλλες ε, συζητήσαμε στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και είχαμε πάει και στην ε, Τουρκία πριν από τα Χριστούγεννα, πήγαμε στο Υπουργείο Άμυνας, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους και στους επαναστάτες από την Συρία και ήταν σαφές ε, το τι θέλει ο Ερντογάν, δηλαδή να εξαλείψει τους τρομοκράτες να μπει δηλαδή στο βόρειο τμήμα του Κουρδιστάν, ε, της Συρίας ε, και να εξαλείψει το PKK, YPG και τους πάντες, όσους πολεμούσαν δηλαδή κατά του ΝΤΑΕΣ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Δεν ακούω πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είπαμε τίποτα για την εισβολή στο Αφρίν. Ε, σιωπή. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτήν την ε, ζώνη ασφαλείας που θέλει να φτιάξει ο Ερντογάν. δεν μπορεί να μπει σε ολόκληρο το Κουρδιστάν, θέλει τουλάχιστον μια τέτοια ζώνη. Μετά αναφέρατε επίσης ότι το Ισλαμικό κρατός ε, κερδίζει έδαφος και ενισχύεται. Και τα ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ε, αυτή τη στιγμή αυτοί ωφελούνται περισσότερο από αυτήν την κατάσταση και η κυρία Λελάνγκ ανέφερε τους ξένους μαχητές ε, που έχουν οι Κούρδοι φυλακισμένους. Έχουμε και άλλους Ευρωπαίους πολίτες ε, στο Ισλαμικό κράτος. Ε, μιλάω για τα παιδιά. Έχουμε παιδιά από την Ευρώπη που ζουν εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα φέρουμε πίσω. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτά τα παιδιά. Thank you, Ms. Valero. And uh, finally from my side, uh, Mr. Και εγώ, τελευταίος ομιλητής. Ένας συνάδελφοι από τη Γεωργία ήρθαν σε επαφή μαζί μου και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αναγνώριση της Συρίας ή μάλλον από τη Συρία, των δύο ε, ε, δαφών ε, ρωσικής κατοχής, Νότιο Σετία και Απχασία. Τι θα κάνει ε, η υπηρεσία σας για τη μία αναγνώριση και έχει ζητήσει από τον Ασάντ να αντιστρέψει αυτή την, ε, την απόφασή του. Έχει έρθει σε επαφή λοιπόν με τη Δαμασκό. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο εκτεταμένα μπορώ. Κάποιες από τις ερωτήσεις πρέπει να πω όμως ε, είναι ερωτηματικά που θέτουμε και εμείς τον εαυτό μας και θα θέλαμε να είχαμε πλήρες απαντήσεις. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα να απαντήσω όμως για τους Κούρδους. Γενικά ακούστηκαν δύο ερωτήματα ουσιαστικά με, που αντιμετώπιζαν το θέμα από διαφορετική σκοπιά. Καταρχάς, η βασική μας ανησυχία ήταν η προστασία των Κούρδων αμάχων και ξεκαθαρίσαμε στην ε, προσέγγιση διαφόρων φορέων ότι η πρώτη εστίαση θα πρέπει να αφορά την ε, προστασία των αμάχων. Κάποιοι από τους ε, ενδιαφερόμενους όμως ε, από τους φορείς ενδιαφέρονται για άλλες κατηγορίες του κουρδικού πληθυσμού. Εμείς και μάλιστα μας είπαν και διάφορους τόπους τους οποίους θέλουν, με τους οποίους τον αντιμετωπίσουν τις άλλες κατηγορίες κουρδικού πληθυσμού. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις επίσης και στα κράτη-μέλη για το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κοινό παρανομαστή στο να προσπαθήσουμε να είμαστε σε επαφή με τους διάφορους ε, φορείς και ενδιαφερόμενους, Τουρκία ειδικά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μονομερείς δράσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν ε, επίπτωση στην ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, στη Συρία. Το θέμα για την ουδέτερη ζώνη. Θα σας δώσω προσωπική απάντηση εδώ, την προσωπική μου άποψη. Για μένα η ουδέτερη ζώνη που πρότεινε η Τουρκία μοιάζει με την ε, ζώνη αποκλιμάκωσης που είχε προτείνει η Ρωσία για άλλες ε, περιοχές ε, της Συρίας και είδαμε πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Είδαμε ότι η τακτική ήταν, αντί να αποκλιμακώσουν, ήταν να κλιμακώσουν σε, ένα επίπεδο τόσο ακραίο που δεν μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω. Επομένως, αναγκαστικά η κατάσταση αποκλιμακωνόταν από αυτό το ακραίο επίπεδο. Και ελπίζω να μην είναι αυτή η μοίρα της ε, συνοριακή περιοχής όπου κατοικούν ε, οι κουρδικοί πληθυσμοί. Υπήρχε μια, υπήρξε μια αναφορά στο Ιντλίμπ. Το Ιντλίμπ όντω έχει καταληφθεί από την Αλνούσρα. Έπρεπε να σταματήσουμε, χρειάστηκε να σταματήσουμε κάποια προγράμματα τα οποία είχαμε εκεί, στο Ιντλίμπ και γύρω από το Ιντλίμπ γιατί είχαμε τους τοπικούς δήμους, τα τοπικά συμβούλια, τα οποία τα έχουν καταλάβει πλέον οι μαχητές του Αλνούσα ή αντίστοιχα, αντίστοιχες ομάδες, ας πούμε. Η κατάσταση είναι μη βιώσιμη. Υπάρχει περίπτωση το καθεστώς λόγω των προβλημάτων αλλού στα βόρεια να εστιάσει να μην, εστιάσει, να μην μπορεί να εστιάσει στο Ιντλίπ. αλλά μπορεί να δώσει έμφαση στο Ιντλίπ το καθεστώς και μπορεί να μπορέσει να το ανακαταλάβει, να μην είναι τόσο δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Ε, τώρα, είχαμε επαφές με τον Ασάτ και τους α, τζιχαντιστές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη, δεδομένου ότι στην αρχή του πολέμου, ο Ασάντ είχε ελευθερώσει διάφορους τζιχαντιστές από τις φυλακές του και ο ίδιος συνεισέφερε τελικά, δημιούργησε μια κατάσταση δύσκολη, επιδεινώθηκε η κατάσταση λόγω της απελευθέρωσης αυτής. Δεν το θέλει αυτό λοιπόν. Τώρα για τη διάσκεψη των Βρυξελών υπάρχουν κάποιες δεσμεύσει. Όταν βλέπουμε τις ανάγκες, ε, οι οποίες δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται, ελπίζουμε ότι οι διεθνείς δωρητές θα μπορέσουν να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με πέρυσι. Σωστά μιλάτε για το γεγονός ότι υπάρχει μια φαιά ζώνη ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και κάποιες μορφές βοήθειας προς ανοικοδόμηση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια και που είναι πολύ προσεκτικοί για το πώς ε, κάνουν τη δουλειά τους και είναι σαφές ότι τα καθαρά ανθρωπιστικά θέματα, ανθρωπιστική βοήθεια και τα κατεπήγοντα είναι αυτά τα οποία ε, μας απασχολούν. Η λογοδοσία είναι ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε. Θα συζητηθεί στην τρίτη διάσκεψη των Βρυξελών και αυτό και έχει συζητηθεί και στο παρελθόν με πάρα πολλέ εκδηλώσει και στην πρώτη διάσκεψη και στη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελών για το θέμα τη λογοδοσία και φέτο επίση θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ένα ερώτημα ακούστηκε επίση ε, για τον ε, ISIS, του Ευρωπαίου πολίτε ε, μέλη του ISIS και τα παιδιά. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών κυρίως αυτό, για το πώ θα αντιμετωπίσουν του δικού του πολίτε. Πιστεύουμε ότι στην περίπτωση των παιδιών τουλάχιστον ε, μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε στη μοίρα τους και ότι μπορούμε να δώσουμε βοήθεια ούτω ώστε να τα επανεντάξουμε σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να ξεπεράσουν τα τραύματα που έχουν ζήσει στη Συρία, στα χέρια και στις περιοχές που κρατούσε ο Άισις. Αυτό είναι όμως ε, αρμοδία των κρατών μελών. Για την αναγνώριση της Συρίας, της Αυχασίας και της Νότιας Οσετίας ε, ήρθαν όντω σε επαφή μαζί μας οι Γεωργιανοί και παρότι οι επαφές μας σε, με τη σφοριακό καθεστώς είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, ήρθαμε και είπαμε ότι κάτι τέτοιο δεν βοηθάει καθόλου, είπαμε στο καθεστώς της Συρίας. Γκράτσι, όπως λέμε και στα Μαλτέζικα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή τύχη στο έργο σας και καλή επιτυχία για την επόμενη διάσκεψη των Βρυξελών που θα οργανώσετε. Συμμετείχα στην τελευταία διάσκεψη και είδα τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Πατή Εκπρόσωπος και πολλοί άλλοι για το θέμα αυτό. Μάλιστα, και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 5, που είναι ένα σημείο με το Ζουάου Βάλε Αλμέιδα. Ε, είναι εδώ ο κύριος Αλμέιδα. Ε, Μένει πως έξω, μπορεί κάποιος να το ελέγξει. He's here. Where is he? Item number five. Σημείο 5. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον πρέσβη Ζωάο Δε Αλμέιδα, πρέσβη της Ευρωπαϊκή Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είμαστε ιδιαίτερω ευτυχείς που παρευρίσκεστε για άλλη μια φορά στην Επιτροπή μας. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για την διοργάνωση μιας επίσκεψης τον προηγούμενο Οκτώβριο για τα μέλη της ΑΦΕ, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Νέα Υόρκη. Ήταν πολύ επιτυχημένη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση επί μία ώρα που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΑ, τον κ. Κουτιέρες. Έχουμε προσκαλέσει και στις 4 Μαρτίου την ε, πρόεδρο της 57ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ε, από το Εκουαδόρ, την κυρία ε, Φερνάντες. Θα ήθελα να σας ακούσουμε την αρχική σας τοποθέτηση για την κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω προσπαθήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια που υπηρετώ σε αυτή τη θέση να επισκέπτομαι την Επιτροπή σας μια φορά το χρόνο. Γνωρίζω ότι μας πιέζει ο χρόνος, έχει πάει και αργά το απόγευμα, επομένω θα προσπαθήσω πολύ τηλεγραφικά να σας εκθέσω τις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις και μετά να ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων που είναι πάντοτε πολύ χρήσιμη. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά ζητήματα, όμως θα ξεκινήσω περιγράφοντας την κατάσταση σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε στο μέσο μιας ιδεολογικής ε, συζήτησης ή και σύγκρουσης. Μια ουσιαστική συζήτηση και δύσκολη συζήτηση. Ανάμεσα σε εκείνους που πιστεύουν ότι στα παγκόσμια προβλήματα πρέπει να βρίσκονται παγκόσμιες απαντήσεις στη βάση κανόνων και μιας πολυμερούς προσέγγισης αφενός και εφετέρου εκείνους που πιστεύουν ότι το πρωταρχικό είναι η εθνική κυριαρχία, είναι το, ο ανταγωνισμός που θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ εθνικών κρατών και ότι τελικά οι λύσεις θα προκύπτουν από την ε, ισορροπία δυνάμεων. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την πρώτη προσέγγιση. Ότι δηλαδή επιθυμούμε ένα διεθνές ε, περιβάλλον που να βασίζεται στους κανόνες, που να ε, προασπίζει τις ε, θεμελιώδες αρχές, το κράτος δικαίου και που να επιδιώκει την συνεργασία, όχι τη σύγκρουση μεταξύ των κρατών και των λαών. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πάντοτε γινόταν, όπως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχει εξυνθεί για λόγους που νομίζω γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Και αυτό είναι το η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Δεν είναι φυσιολογική και οι εποχές που διανύουμε. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, μια περίοδο όπου έχουμε ανατροπή του πολυμερούς συστήματος, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η δικιά μου δουλειά, το δικό μου έργο στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι και ο Οργανισμό των Εθνών είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Έχουμε για πρώτη φορά έναν πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό είναι, ε, με κάνει πολύ ευτυχή, μιας και έρχεται και από την χώρα μου, από την Πορτογάλος, αλλά είμαι ακόμα πιο ευτυχής επειδή είναι Ευρωπαίος και ο οποίος προσπαθεί να εφαρμόσει ε, Φιλόδοξε μεταρρυθμίσεις με εκείνου που θέλουν να τι υποστηρίξουν. Έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Το 2019 θα εφαρμοστούν διάφορε σημαντικέ πρωτοβουλίε και ιδέε που είχε αναπτύξει. Κατά την άποψή μου, αυτή η μεταρρύθμιση προχωράει ικανοποιητικά, δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει κατά την άποψή μου τον Γενικό Γραμματέα σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί για να υπεραμεινθούμε τις πολυμερούς προσέγγισης. Για να τα καταφέρουμε να συμβεί αυτό, να παραμείνει ο ΙΕ στο κέντρο μιας πολυμερούς προσέγγισης των διεθνών προβλημάτων, πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση του για να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις κουτιέρες είναι πολύ σημαντικέ. Και είναι ένα θέμα που θα ε, έλθει στο 2019, θα, θα αναδειχθεί, που θα είναι δύσκολο, είναι ο προϋπολογισμός του ΟΗΕ. Γνωρίζω ότι το, γνωρίζετε το θέμα, αλλά θα το επαναλάβω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει περίπου το 1 τρίτο τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ. Το 1 τρίτο. Περίπου το 30% για να είμαστε ακριβεί. Έρχεται από του φορολογουμένου των κρατών μελών, τους, των, ε, που εσεί εκπροσωπείτε εδώ. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Εκτό αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει τι συνεισφορέ τη πλήρω, εγκαίρω και δεν σταματάει να πληρώνει τα χρέη της. Εάν το ίδιο έπραταν και οι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του κόσμου, δεν θα βρισκόταν ο ΙΕ στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα, την οποία θα εκθέσει ο Γενικό Γραμματέα και θα αναζητηθούν λύσει. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για την συστηματική και τακτική υποστήριξη του ε, προπολογισμού του ΟΗΕ το οποίο οφείλεται και σε εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ω αρχική ελέγχου του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση στα κράτη-μέλη. Θα έλεγα ότι γενικά ε, εγώ είμαι έτσι ένας αισιόδοξο άνθρωπο. άνθρωπος, με γνωρίζουν το γνωρίζουν, αλλά θα έλεγα ότι γενικότερα είμαι ευτυχή ω πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε αποτέλεσμα στον ΟΗΕ. Θα σα δώσω ορισμένα παραδείγματα. Καταφέρουμε να είμαστε ενωμένοι και στο 93, 94, 95% των περιπτώσεων να ψηφίζουμε ε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντεταγμένα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά καταφέρνουμε να, να τις συζητούμε, οργανωνόμαστε και καταλήγουμε σε κοινέ θέσεις τις οποίες προσπίζουμε στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό και η ομάδα μου και πιστεύω και όλοι οι πρέσβεις των 28 ε, κρατών μελών της Ένωσης στη Νέα Υόρκη είναι περήφανοι γι' αυτό. Να σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα. Είναι η στάση μας στο εσωτερικό του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει πέντε μέλη μόνιμα και μετά δέκα ε, ε, μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Αυτή τη στιγμή είμαστε 8 από τους 15, 5 και 3. Αλλάζουν αυτοί οι αριθμοί των εκλεγμένων φυσικά και τίθεται πάντα το, ερώτημα εάν θα έχουμε μέγιστο αντίκτυπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας εάν συντονιζόμαστε αυτά τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται. Και στον τομέα αυτό θα με χαρά σας ανακοινώνω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα με το οποίο η δική μου η ομάδα φροντίζουμε έτσι ώστε όλες, όλα τα κράτη που είναι μέλη και στο Συμβούλιο ασφάλεια του ΟΗΕ και είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν την ίδια θέση. Με κάποιε παραλλαγέ, φυσικά, αλλά με την ίδια θέση. Και μια, έναν αντίστοιχο συντονισμό προσπαθούμε να πετύχουμε και σε όργανα εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας. Γι' αυτό θα το έχετε διαπιστώσει και στον τύπο, ότι οποτεδήποτε έχουμε, γιατί δεν συμβαίνει πάντοτε αλλά αυτό, αλλά οποτεδήποτε έχουμε μια κοινή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται μια κοινή δήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ένας από τους πρέσβεις θα εκφωνήσει αυτή την κοινή θέση. Εκφωνεί αυτή την κοινή θέση. Το έχουμε κάνει για παράδειγμα σε ζητήματα όπως κλιματική αλλαγή, η Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκπροσωπονώ εγώ όταν έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό έχοντας κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλήσω στο Συμβούλιο ε, Ασφαλείας του ΟΗΕ ως πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και οι πρέσβεις των κρατών παίρνουν το λόγο και ουσιαστικά εκφράζουν την ίδια θέση το οποίο, ε, το οποίο δείχνει μάλλον ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινή και ενιαία έναντι των πολιτών και του τύπου. Αυτό είναι ε, μια πολύ σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών. Όμως, έχω ένα σημαντικό μήνυμα προς εσάς και το οποίο πανέρχομαι, που είναι ε, το να γνωρίζουμε ότι καταφέρνουμε να έχουμε αποτελέσματα όταν είμαστε ενωμένοι. Δεν καταφέρνουμε να έχουμε και τόσο πολλά αποτελέσματα όταν είμαστε διχασμένοι. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο προσπαθώ να μεταφέρω πάντοτε και στους ε, στον κύριο Μακάλιστερ, στου συναδέλφου σας, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μα επισκέπτονται στη Νέα Υόρκη, αλλά είναι σημαντικό να το πούμε και εδώ, να το πω απευθεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση είναι σημαντικό να το ε, μεταφέρετε εσεί και στου πολίτε, σα μια και πλησιάζουν και οι ευρωεκλογέ. Ο κόσμο μα σήμερα είναι περίπλοκος, έχουμε διαρκώ νέε απειλέ, έχουμε εξελίξεις, ακόμα και συμμάχους που τους θεωρούσαμε σίγουρους δεν μπορούμε πια να τους θεωρούμε, έχουμε αμφισβητήσεις. Εν ώψη λοιπόν και των ευρωεκλογών δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τη διεθνή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πόσο σημαντικό είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες να υποφελούνται από αυτή την κρίσιμη μάζα που δημιουργείται όταν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται μεταξύ τους που είναι πολύ σημαντικότερη από τι προσπάθειε που θα μπορούσε να κάνει καθένα του ξεχωριστά. Ελπίζω η συζήτηση που θα γίνει εν ώψη των ευρωεκλογών να μην περιοριστεί μονάχα στα εσωτερικά μα ζητήματα και στα ζητήματα του κάθε κράτου μέλους, αλλά θα έχουμε και να έχουμε και μια συζήτηση για τον παγκόσμιο ρόλο που πρέπει να παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι στο ζήτημα της σχέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΕΕ πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ε, χαρά να συνεργαστώ μαζί σας και με τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ, αλλά και από, με άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεματικές αποστολές. Με μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε, σας ενημερώνουμε και θα έλεγα ότι προσπαθώ να ενθαρρύνω τις ε, επισκέψεις από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο, στη Βάσιγκτον όταν ήμουν. Πολύ συχνά είχα την ευκαιρία τον κύριο Μπρόκ που μόλις μπήκε στην αίθουσα να τον φιλοξενήσω με την ιδιότητα του τότε ως πρόεδρο της ΑΦΕΤ και αντιστοίχω τώρα το ίδιο πράγμα με τον κύριο Μακάλιστα και αντιστοίχω και με άλλου ε, εκπροσώπου ε, των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί μπορείτε εσεί να πείτε ω ε, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου πράγματα που εγώ ίσω να μην μπορώ να πω και με αυτόν τον τρόπο να τονίσετε τι θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το πολυμερή προσέγγιση στα διεθνή προβλήματα και, τις μια προσέγγιση που βασίζεται σε θεμελιώδει αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζωάου Βάλεντε Αλμέιντα. Έχουμε 35-40 λεπτά για ανταλλαγή απόψεων. Μου ζήτησαν να μιλήσουν οι εξή. Ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτού του τέσσερι. Ο κύριο Αλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθε, ε, Ζουάου Βάλεδε Αλμέιδα. Καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνει στα Ηνωμένα Έθνη τα τελευταία χρόνια, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε πριν έρθεις εσύ ε, ψήφιζαν 60% προς τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ τώρα έχουμε τεράστια πρόοδο με την έλευσή σου. Θα ήθελα ο πρέσβης μα στη Νέα Υόρκη, ο θαυμάσιος αυτός πρέσβης στη Νέα Υόρκη, να μας, να μας εξηγήσει τι συνέβη ε, το Σάββατο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την βασική συζήτηση που έγινε Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχει προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική. Ε, ε, το Brexit, ε, το Trump έφερε η τέταρτη αυτή συνεδρία, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τη δημαγωγία. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν να γίνουν εργαλείο παγίωσης της δημοκρατίας ή θα εδραιώσουν καθεστώτα όπως το κινέζικο. Θέλουμε νέα αρχιτεκτονική παγκόσμια, νέα στρατηγική παγκόσμια, διερωτώ με αν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προκαλέσατε, σκέφτονται αυτό το θέμα και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στις ε, εξελίξεις αυτές. Αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Νάτσο Σαλαφράγκα. Και τώρα πάμε στον κύριο Χόιντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Αλμέιδα, Πάντα με χαρά σας ε, υποδεχόμαστε, είτε εδώ είτε στη Νέα Υόρκη. Ε, μόνιμο, μόνιμη φιγούρα, μόνιμος ομιλητής ε, είσαστε τα χρόνια αυτά. Δύο ρωτήσεις. Καταρχάς, ο κύριος Καν μόλις έφυγε, ο κύριος Καν, αφορά το Brexit όμως. Αναφέρατε για πρώτη φορά, νομίζω, άμεσα και ρητά την ε, φοβερή αυτή ομοφωνία που δείχνουν τα ευρωπαϊκά κράτη του Συμβουλίου Αυσταλίας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Έτσι, αραγές μέτωπο εκεί. Τι θα συμβεί. Α, για την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στην ε, Νέα Υόρκη το συζητήσαμε. Τι θα γίνει αν το Brexit ε, οδηγήσει σε no deal, καμία συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει διαφορά εάν έχουμε συμφωνία ή αν δεν έχουμε συμφωνία για τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή είναι μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το χρήμα. Ε, είπατε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το 1 τρίτο όλων των χρηματικών αναγκών, καλύπτει το 1 τρίτο των χρηματικών αναγκών του ΟΗΕ. Εάν αναπατώμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Το ίδιο σωστό, όχι, περίπου το ίδιο λέει ο κύριος Αλμέιδα. Ακούσατε πάντως πρόσφατα τίποτα για τη συνεισφορά των Αμερικανών που θα περικοπεί σημαντικά, θυμολογείτε. Ή είναι οι φήμες που ακούγονται με κάθε νέα αμερικανική κυβέρνηση που θεωρούν τον ΟΗΕ γραφειοκρατικό, επαχθή, ε, και πολύ ακριβή και πολύ ακριβώς οργάνωση. Ευχαριστώ κύριε Φόιντ. Κύριε Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και κύριε Πρέσβη που ήρθατε και πάλι να μοιραστείτε μαζί, σας, μαζί μας την ανάλυση σας. Κάθε χρόνο έχουμε ένα ψήφισμα και εκεί πέρα λέμε ότι ζητάμε μια μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Φέτος τον Ιούλιο ε, ζητήσαμε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση αυτή μέσω της ε, μείωσης ε, του δικαιώματος του ΒΕΤΟ, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου. Τώρα έχουμε πέντε μέλη μόνιμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά φαίνεται ότι οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση είναι ακόμα μπλοκαρισμένες τι θα μπορούσε να βοηθήσει να αλλάξει η κατάσταση. Και μετά για την Ιεμένη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ακρόαση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κατάσταση στη χώρα αυτή και όλοι οι ειδικοί επανειλημμένως ζήτησαν απαγόρευση της εξαγωγής όπλων και σε μέλη της Σαουδαραβικής Συμμαχίας. Βεβαίω, κάποια κρατημέλη έχουν αναστείλει τις εξαγωγές στη Σαουδική Αραβία η Αμερικανική Γερουσία πέρασε μια νομοθεσία που λέει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο. Βλέπετε εσείς ε, κάποια δυνατότητα να υπάρξει απαγόρευση εξαγωγών όπλων προς την Ιεμένη. Σας ευχαριστώ Χέλμουντ Σόλτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρέσβη και χαίρομαι που είστε εδώ. Αναφέρατε πολλά τέτοια ζητήματα. Αλλά με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο στις ΗΠΑ, πώς θα χαρακτηρίζατε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να λάβουν περαιτέρω ενεργά ναι, μέρους ε, στη μεταρρύθμιση του συστήματος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ή υπάρχει πάντα πίεση από την Ουάσιγκτον ε, για μείωση της συνεισφοράς των ΙΠΑ και βεβαίω και των ευθυνών του στι διεθνεί Δεύτερον, έχουμε συζητήσει τα ζητήματα κλιματική αλλαγή, Παρίσι κτλ. Τα νέα αυτά θέματα λοιπόν. Πώς επηρεάζουν ακριβώς ε, την ε, δουλειά του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πώς ε, βλέπετε τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ δύο συνάδελφοι ακόμα, Εντουάρντ Κούκαν και μετά η Γκόμες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Πρέσβη όλοι εκτιμούμε ιδιαιτέρως ε, τη δουλειά που κάνετε και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι. Πριν από λίγο χαιρετήσαμε τον Σταύρο Λαμπερνίδη, ο οποίος πηγαίνει στην Ουάσιγκτον επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ένωσης. Οπότε η ερώτησή μου είναι παρόμοια με αυτά τα οποία είπε ο κ. Σόλτς. Πώς ε, θα, αξιολογούσατε την πολιτική των ΙΠΑ για τον ΟΗΕ. Αντιλαμβάνομαι ότι θα στείλουν και μια νέα πρέσβυρα αναμένει την ακρόασή της. Είναι απρόβλεπτος ο Λευκός Σύκο. Πώς τα βλέπετε εκεί στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ ποτέ δεν ήταν πολύ δημοφιλής της ΙΠΑ. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Κατόπιν ε, για τις ε, ρωσικές δραστηριότητες και την συμπεριφορά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Or Αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια επαφή συνεργασία ή υποψία συνεργασίας με τη Ρωσία ή είναι παντελώς αδύνατον. Καλή τύχη εύχομαι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποια σχέδια για το Brexit και δεδομένου του ότι ξεκινάει η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς εμάς ε, αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια αναβαθμισμένη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα λάξ στην έδρα της Γαλλίας. Δεύτερη ερώτηση. Είχαμε ήδη μια δύσκολη συζήτηση για τη Βενεζουέλα. Προς τα που πάμε. Προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο ή θερμό πόλεμο. Δεδομένου του ότι η Ρωσία έχει βομβαρδιστικά ε, ή καν αναφέρουν πυρηνικά όπλα στη Βενεζουέλα. Μετά. Ανθρώπινα δικαιώματα και ο ΙΕ ε, μόλις επιστρέψαμε κάποιοι από εμά από την ε, Νικαράγουα, από την ηγεσία του Χαμόνα Ρέγγι, όπου το... από όπου απελάθηκε η εκπρόσωπος του είπα του ΙΕ για ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και... Βεβαίω δεν ακούει πολλά κανεί εκτό τη χώρα και λένε εντάξει, γιατί κάνει βαβούρα ο ΙΕ τι κάνει ο ΙΕ παραδείγματο χάρη ε, για ζητήματα όπως η δολοφονία του Κασόγκη. Ε, παραδείγματο χάρη μιλάει πάρα πολύ καλά για τη συνεργασία που υπάρχει με την ύπατη αρμοστία του ΙΕ ε, για τους πρόσφυγες και αυτό βέβαια επηρεάζει την κατάσταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν αλλά δεν ακούμε πολλά πράγματα από εκεί. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτές τις παρατηρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση στον ΟΗΕ σε σχέση με την ε, κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, μιας και διαγράφεται σιγά σιγά και μια εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου από, τον, ε, από το φθινόπωρο και τι έχει συμβεί σχετικά. ο κύριο Βάλτε Αλμέιδα. Είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσαμε να συζητούμε όλο το απόγευμα, αλλά μάλλον θα έχετε άλλα σχέδια. Επομένω, θα προσπαθήσω συνοπτικά να απαντήσω στι ερωτήσει σα και ίσω ομαδοποιώντα ορισμένε από αυτέ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για τα καλά σα λόγια. Θα τα μεταφέρω και στου συνεργάτε μου. Όταν μιλώ για του συνεργάτε μου, είναι οι 28 πρέσβει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ και με του οποίου έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Για το ζήτημα της Βενεζουέλας. Δεν παρευρέθη στην ε, συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα αυτό, γιατί βρισκόμουν καθοδόν για τις Βρυξέλλες, αλλά ενημερώθηκα και γνωρίζουμε όλοι ότι η συζήτηση ήταν δύσκολη και ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Για την ακρίβεια έγινε συζήτηση για το εάν θα έπρεπε να γίνει συζήτηση. Επ' αυτής η συζήτηση θα έλεγα ότι κερδίσαμε επειδή έγινε συζήτηση και τουλάχιστον φάνηκε ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στη, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί τις εξελίξεις προσεκτικά, το γνωρίζω, και σε μεγάλο βαθμό προσπαθεί να βρει μια λύση η οποία να συγκλίνει με τις προθέσεις της, ε, τις, τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να επιλύσει την κατάσταση. Όμως είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε σχέση με την ε, νομιμοποίηση που έχει ή δεν έχει ο πρόεδρος Μαδούρο και καθώς επίσης ε, την υποστήριξή μας στους μηχανισμούς που προβλέπει το Σύνταγμα για να λυθεί αυτή η κρίση. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι για το θέματα που θέτει ο κ. Σαλαφράγκα και η κυρία Γκόμε, ε, που είναι η ανησυχία να μην υπάρξει ένας εκτροχιασμός της κατάστασης που θα έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις για τους ε, πολίτες της Σε Αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η κυρία Μογκερίνη τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες. Έχει επικοινωνήσει με διάφορους ηγέτες ε, στην περιοχή, με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ, προσπαθώντας να βρεθούν κάποιες λύσεις πολιτικές, κάποια βήματα που θα οδηγήσουν σε πολιτικές λύσεις για το θέμα αυτό. Όμως γνωρίζουμε όλοι ε, ότι η ανησυχία είναι ο εκτροχιασμός. Στην Ιαϊόρκη συμβουλευόμαστε όλους τους εταίρους μας, όμως έχουμε απέναντί μας, και πρέπει να το πω αυτό, χώρες κάτι τα οποία θεωρούν ότι εδώ πρόκειται για μια παρέμβαση στα εσωτερικά μιας κυριαρχής χώρας. Και ερχόμαστε εδώ στην πρώτη παρατήρηση που έκανα για την ε, συζήτηση, για την διαμάχη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο ανάμεσα σε εκείνους που πίζουν την ε, πολυμερή προσέγγιση στα διεθνή προβλήματα και τους άλλους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο άμεσο μέλλον και πώς θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Αναφερθήκατε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τι τελικά αντίκτυπο είχαν αυτά στη δημοκρατία και στις διεθνείς σχέσεις. Θα έλεγα ότι έχουμε αντιληφθεί τη σημασία αυτών των εξελίξεων και θα σας δώσω δύο παραδείγματα και ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και η κυρία Μογκερίνη έχουν δημιουργήσει task force, ομάδε εργασία για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, στι οποίε συμμετέχουν εμπειρογνώμονε με πολύ ψηλά προσόντα και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Στόχο αυτών των ομάδων είναι κοινό. Να αντιληφθούμε καλύτερα ποιες ε, θετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι επαναστάσεις τεχνολογικές αλλά επίσης να αντιληφθούμε και τις διάφορε παγίδες, τους διάφορους κινδύνους που εγκυμονούν. Είδαμε, για παράδειγμα, τη χρήση της τεχνητή νοημοσύνης, ε, την πιθανότητα μάλλον να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο να έχουμε όπλα τόσο έξυπνα, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών στο μέλλον, που να αποφασίζουν μόνο του πόσοι θα ε, σκοτωθούν. Ε, Αυτέ είναι εξελίξει τις οποίε σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να, να παραμείνουν αδρανή τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει εντοπιστεί ω μία από τι σημαντικέ προτεραιότητε για τον ΟΗΕ από την πλευρά του Γενικού Γραμματεία για το 2019 και επίση θα έλεγα ότι και για την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Μογκερίνη ε, θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλή προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Νομίζω σε αυτό τουλάχιστον όλοι συμφωνούμε. Για το ζήτημα του Brexit μου ετέθησαν διάφορα ερωτήματα δεν είναι ένα ζήτημα που γνωρίζω και είναι ένα ζήτημα πολύ περίπλοκο και πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα ήταν ε, ορθό εκ μέρου μου να υπερβώ τι αρμοδιότητέ μου και να κάνω κάποιο σχόλιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παρακολουθούμε τι εξελίξει στην Ευρώπη προσεκτικά και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα μετά το Brexit. Επίσης μας ενδιαφέρει η μεταβατική περίοδος, αλλά επίσης μας ενδιαφέρει και η μελλοντική σχέση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα ζήτημα ιδιαίτερο ενδιαφέροντος ε, στη Νέα Υόρκη, φυσικά, είναι ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι αμέσω μετά τον Brexit το, οι θέσει του Ηνωμένου Βασιλείου θα αλλάξουν άρδιν σε σχέση με αυτές που μέχρι τώρα ε, υποστήριζε. Άρα πιστεύουμε ότι μέχρι στιγμή, τις περισσότερες των περιπτώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούσε με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φανταζόμαστε ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον. Ότι δεν θα δούμε ξαφνικά μεγάλες διαφορές. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι είναι απολύτω φυσιολογικό να αναζητήσουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit για ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, εμπορίου, ε, διεθνών σχέσεων κτλ. Ε, από την πλευρά μου, όπω παρακολουθώ εγώ τα πράγματα από τη Νέα Υόρκη, μου φαίνεται το φυσιολογικό, το προφανέ. Βεβαίω, επίση προφανέ είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένω υπάρχουν διαφορέ. Υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα σε ένα μέλο και ένα μη μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πρέπει να βρούμε τρόπου με του οποίου η συνεργασία θα είναι στενή, σεβόμενη όμω ταυτόχρονα το γεγονό ότι η χώρα αυτή δεν είναι πια μέλο. Για το ερώτημα που μου έθεσε ο κύριο Φρόιντ για την πιθανότητα εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρί τη συμφωνία. Και πάλι δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο, είναι το ζήτημα ευαίσθητο. Θα δούμε όταν έρθει αυτή η στιγμή πώ θα οργανωθούμε. Βεβαίω, η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία συμφωνώ και εγώ και την επαναλαμβάνω είναι ότι θα είναι λάθο να υπάρξει έξοδο χωρί συμφωνία και επίση θα, δημιουργη... θα είναι πιο δύσκολο να υπάρξει συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο αν αποχωρήσει χωρί συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει και μία μεταβατική περίοδο, η οποία θα μα διευκολύνει. Ενώ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, τα πράγματα σίγουρα θα περιπλακούν αλλά βλέποντα και κάνοντα θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει. Μιλώντα τώρα για το μέλλον του Συμβουλίου Ασφαλεία μετά τον Brexit. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναφέρθηκα και το οποίο σχετίζεται και με, τις μεταρρυθ... τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι στο ίδιο μήκο κύματο, δεν συμφωνούν για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και να ένας τομέας στον οποίο δεν συμφωνούμε, γι' αυτό και δεν μπορώ να πω ότι συμφωνούμε στο 100% των θεμάτων που συζητούνται στη Νέα Υόρκη. Όχι, εδώ έχουμε ξεχωριστές θέσεις κρατών μελών διαφορετικές. Και όταν μιλώ για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλεία, μιλώ για την πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμό των μελών του, να αλλάξει ο τρόπο λειτουργία του, το βέτο κτλ. Ε, δεν μπορώ να εκφράσω εγώ μια θέση δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη εδώ έχουν διαφορετικέ θέσει μεταξύ του. Για το ζήτημα όμω του να περιοριστεί το δικαίωμα χρήση του βέτο όταν έχουμε περιπτώσει γενοκτονία, που αναφέρατε, είναι μια συζήτηση στην οποία έχουν συμμετάσχει κάποια κράτη-μέλη. Δεν έχει κοινή θέση στην Ονισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό, το παρακολουθεί. Ε, αυτό που διαπιστώνω εγώ στην Νέα Υόρκη είναι να γίνεται ένα ζωντανό και έντονο διάλογο για ένα θέμα σημαντικό και το παρακολουθώ ω παρατηρητή. Και διαπιστώνω ταυτόχρονα ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλεία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από όλο και περισσότερα κράτη-μέλη τη Ένωση. Βεβαίω αυτό θέτει και ένα ουσιαστικό, όχι απλώ ακοδημαϊκό ερώτημα, είναι αν μπορούν να γίνονται βηματικά μικρέ μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς να υπάρχει μια συνολική συμφωνία για μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Απαντώ εν μέρη στην κυρία Λόχμπιλα και θα ήθελα να την ευχαριστήσω με την ευκαιρία και εκείνη και, ε, στους συναδέλφους, συναδέλφους της στην ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε συνεργασία τα τελευταία χρόνια πολύ καλή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την, ε, το χρόνο και την ενέργεια και το έργο που έχετε επενδύσει και ελπίζω να συνεχίσει αυτή η συνεργασία και αυτό το έργο και με τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έλεγα ότι αυτή η θητεία του, κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε μια μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του Κοινοβουλίου να εμπλακεί και να συνεργάζεται και να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον ΟΗΕ. Με ρωτήσατε επίση και για την Ιεμένη. Αναφέρθηκα στο ζήτημα τη πολιτική βούληση ε, των εξελίξεων. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια ορμή για πολλούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους και η δολοφονία Κασόγκη, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκόμες. Διαπιστώνω ότι ο Γενικός Γραμματέας θέλει να αξιοποιήσει αυτή την εξέλιξη, αυτή την όθηση. Έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Έχει αποστείλει, για παράδειγμα, μια αποστολή στην Ιεμένη με ουσιαστική εντολή αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής καταστροφής, γιατί αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η όφηση, έτσι ώστε να φτάσουμε τελικά σε μια πολιτική ε, διαδικασία, διαδικασία πολιτικής επίλυσης του προβλήματος δηλαδή. Τώρα αν αυτό συμπεριλαμβάνει και την απαγόρευση πώληση όπλων, δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί υπάρχουν, επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ο ειδικό ανταποκριτή ε, του ε, Γενικού ο κ. Ρίφιτ, απολαμβάνει τη υποστήριξη τη Γενική Συνέλευση και τη εμπιστοσύνη του Γενικού Γραμματέα. Την ίδια εμπιστοσύνη έχει, έχει και από εμά. Για τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Πράγματι ήταν το ζήτημα τη εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι Ηνωμένε Πολιτείε αυτό που με απασχολούσε πριν μεταβώ στη Νέα Υόρκη. Έχω ζήσει και 9 χρόνια στι ΗΠΑ, πώ να μην κάνω σχόλιο. Βέβαια, είναι ο νέο μα πρέσβη, ο κ. Λαμπρινίδη, αυτό που θα πρέπει στο μέλλον να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Το μόνο λοιπόν που θα κάνω είναι να σα δώσω μια, να σας κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τι εμπειρίε που έχω αποκομίσει στον ΟΗΕ. Έχω δει διάφορε κυβερνήσει των Ηνωμένων Πολιτειών πάντοτε να λαμβάνουν επικριτικές θέσεις έναντι του ΟΗΕ. μια σημαντική διαφοροποίηση ίσως να υπήρξε κατά τη δεύτερη θητεία Ομπάμα. Αλλά κατά τα άλλα θα έλεγα ότι όλες οι κυβερνήσεις των Πολιτειών επικρίνουν τον ΟΓΕ για οικονομικούς λόγους, για λόγους αρχής. Και επομένω, νομίζω κανένα δεν εκπλήσεται όταν διαπιστώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθυγραμμίζονται με τον ΟΗΕ ε, πάντοτε με μια επικριτική διάκριση. Προσεγγίζουμε μάλλον τον με μια επικριτική διάθεση. Όμως αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν αμφισβητηθεί οι θεμελιώδεις αρχές η θεμελιώδης διάρθρωση του πολυμερούς διεθνού συστήματος από τον πρόεδρο Τραμπ. Και γι' αυτό έθεσα έτσι το ζήτημα στην αρχή της παρέμβασής μου, ότι η διαμάχη και ο διάλογος που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για το τι σημαίνει πολυμερές ε, διεθνές σύστημα πιστεύω ότι η προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε εμείς εδώ είναι μια προσέγγιση διπλωματική, συζήτηση και διαρκή. Υπάρχει επίση και η οικονομική διάσταση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ανασυχεί το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποφασίσει να μην πληρώσουν το 28% που τους αναλογεί για τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Δεν θέλουν να πληρώσουν πάνω από 25% το οποίο σημαίνει ότι κάθε χρόνο, σε αιτήσια βάση, το 3% της ε, συνεισφοράς της οικονομικής που θα περίμενε κανείς από τις Ηνωμένες ε, Πολιτείες δεν έρχεται. Και αυξάνονται τα χρέη. Και δεδομένου μάλιστα ότι η διάρθρωση του προϋπολογισμού του ΟΗΕ είναι αυστηρή, δεν έχει το δικαίωμα ο Γενικό Γραμματέα να μετακινεί κονδύλια από τον ένα τίτλο του προπολογισμού στον άλλον. Επομένω, το ζήτημα δεν μπορεί να επιληθεί στο σε εσωτερικό επίπεδο από το Γενικό Γραμματέα. Και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησε στρεβλώσεις ε, περίεργες, ε, για παράδειγμα στον αριθμό των στρατευμάτων που συνεισφέρουν κάποια κράτη. Γιατί δεν μιλούμε για απλώ για συνεισφορά οικονομική, μιλούμε για συνεισφορά σε ανθρώπου, σε στρατιώτε, οι οποίοι σε ορισμένε περιπτώσει σκοτώνονται Και αυτή η κατάσταση με την μη κάλυψη των υποχρεώσεων των οικονομικών των ΗΠΑ για τι ρευστικέ αποστολέ έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρέη από τον ΟΗΕ προ κράτη, τα οποία θα αντιστοιχούσαν σε 200 χρόνια συνδρομών του κράτους αυτού προς τον ΟΗΕ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ ανησυχητική, ανησυχεί και το Γενικό Γραμματέα και εμάς και μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη μας πληρώνουν τις συνεισφορές τους με βάση τους κανόνες, στην ώρα τους και για όλους τους σκοπούς. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια άλλα κράτη τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Εδώ είναι λοιπόν μια συζήτηση η οποία πρέπει να τεθεί, θα τεθεί από τον Γενικό Γραμματέα. Τώρα για την νέα πρέσβη του Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, τον, την περιμένουμε και όπως πάντοτε θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνεργασία, συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επιδιώξουμε να, έχουμε, να βρίσκουμε ε, τα κοινά σημεία, της τα σημεία που είναι πολλά υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε και με αυτή την Αμερικανική κυβέρνηση και θα προσπαθήσουμε να τους αξιοποιήσουμε στο επίκρο. Κλείνω. Για την κλιματική αλλαγή, κύριε Σόλτς. Αναφέρθηκα στις προτεραιότητες του Γενικού Γραμματέα, είναι η κλιματική αλλαγή μία από αυτές, γιατί διαπιστώνουμε ότι εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή πολύ πιο γρήγορα από ότι εμείς αντιποκρινόμαστε σε αυτήν. Ε, ε, το επαναβεβαιώσαμε στη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο, στη σύνοδο του Κατόβιτσε τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από αυτά που περιμέναμε, αυτό μας ενθαρρύνει. Αλλά συνεχίζουν να πρέπει να γίνουν πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώ ηγείται αυτή τις προσπάθειες Και επίσης την τελευταία εβδομάδα συζητήθηκε το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο Ασφαλείας Παλιά, όταν έφτασα εγώ στην ε, Νέα Υόρκη, υπήρχαν κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα οποία αρνούνταν να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρούσαν ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχει αλλάξει αυτό πια. Θα έλεγα ότι είναι πλέον τακτικό θέμα συζήτηση. και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στι παραμβάσει των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως εάν προχωρήσει η κλιματική αλλαγή όπως πάει, θα υπάρχει αντίκτυπος σε ζητήματα ασφαλείας. Θα μεταναστεύει ο κόσμος μαζικά για αυτόν τον λόγο. Εκατομμύρια εκατομμυρίων θα μετακινούνται και αυτό μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε καλά κάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας και το κοιτάει και ο Γενικός Γραμματέας και το 2019 να μένουμε περαιτέρω πρόοδο. Όσον αφορά την συνεργασία με την Ρωσία, έφυγε ο κύριος Κούκαν. Ε, η Ρωσία είναι βεβαίω μια χώρα αναντικατάστατη, όπως τα έλεγαν οι Γάλλοι. Δεν μπορούμε και να την αποφύγουμε στον ΟΗΕ για τους προφανείς ε, λόγους. Ε, μόνιμο μέλο του, του Συμβουλίου ασφαλεία. Επενδύουν πολλά, έχουν καλούς διπλωμάτες. Ε, βεβαίω είμαστε σε επαφή σε τακτική βάση. Πρέπει να πω ότι τις περισσότερες φορές είμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα για διαφορετικούς λόγους. Όποτε μπορούμε και υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε. Βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε με τους Ρώσους φίλους μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Τελευταία πρέπει να αναγνωρίσω. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Άννα ε, βεβαίως ε, έκανε μια πολύ σωστή ερώτηση. Είναι ζωτικό κομμάτι του ΟΗΕ. Το άλλο θέμα το οποίο αναφέρατε βεβαίω είναι ζήτημα της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Μισελ Μπασλέ δεν χρειάζεται νομίζω να την επενέσω εγώ και ο Γενικός Γραμματέας αποδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα όπως και εμείς. Ε, νομίζω λοιπόν πως ε, μόλις η κυρία Μπασλέ εξοικειωθεί με το θέμα θα πρέπει ακριβώς ε, να τις δώσουμε το απαραίτητο περιθώριο. Ε, πράγματι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ικαράγουα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, χωρίς αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι κάπως ανησυχητική και από την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρος πως η κυρία Μπασλέ και ο Γενικός Γραμματέας αποδίδουν την κατάλληλη σημασία. Τελευταία ερώτηση από τον πρόεδρο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, το είχαμε συζητήσει μερικές φορές ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και οφείλω να πω ότι δεν έχω δει σημαντική πρόοδο ε, στο θέμα αυτό, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουμε να ε, συνεργαζόμαστε με τη Σερβία, το Κοσφοπέδιο, η κυρία Μογκερίνη παίζει κέριο ρόλο στην διευκόλυνση του διαλόγου και στη Νέα Υόρκη αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου που θα μας ε, βοηθήσει να έχουμε κάποια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θα τελειώσω λοιπόν ευχαριστώντας σας ακόμη μια φορά για την φιλοξενία σας, ε, για τις δεσμεύσεις σας. Είναι τελευταία φορά που έρχομαι ενώπιον της Επιτροπής σας ως των ΙΕ και έχω την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές όσοι είστε ξανά υποψήφοι και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την καλή συνεργασία που είχαμε στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα τελευταία 8 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, colleagues. Any further questions, comments from your side? Όλοι συνάδελφοι. Όχι. Ευχαριστώ Ζουάου που ήρθε στην Επιτροπή μας. Καλή τύχη. Και τώρα. Έχουμε 7 λεπτά διάλειμμα και μετά θα έρθει εδώ ο κύριος Χωσέ Βαλένθια. Ο κύριος Χαουρέγγι θέλει να έρθει εδώ δίπλα μου. So. Ladies Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Προχωρώντα στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Χωσέ Βαλένσια, Υπουργό Εξωτερικών και Ανθρώπινη Κινητικότητα του Εσημερινού, ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του προηγουμένου έτους. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα Ισπανικά. Στην ε, συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να κάνω ορισμένες ε, ναρκτήρε παρατηρήσεις πριν σας δώσω το λόγο. Θεωρώ ότι η επισκεψή σας καταδεικνύει την προσπάθεια που κάνει η τρέχουσα κυβέρνηση του σημερινού να ανοιχθεί προ τον κόσμο και να συνεργαστεί με άλλες χώρες, αλλά κράτη του κόσμου για τα σημαντικά παγκόσμια προβλήματα. Καλωσορίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι ο σημερινό είναι μια χώρα πολύ σημαντική για τη σταθερότητα στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι το Εκουαδόρ έχει επηρεαστεί σημαντικά από την προσφυγική κρίση της Βενεζουέλα. Έχετε επιδείξει εξαιρετική ε, φιλοξενία και έχετε αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη εισρωή προσφύγων. Ταυτόχρονα βέβαια η κατάσταση και η κρίση στη Βενεζουέλα φαίνεται να επιδεινώνεται καθημερινά ε, μετά την ανανέωση της θητείας για άλλα 6 χρόνια του Πρόεδρου Μαδούρο. Ελπίζω να συζητήσουμε το, όχι μόνο το ζήτημα της κατάστασης στη Βενεζουέλα, αλλά επίσης και της κατάστασης στην Κολομβία. Έχει παίξει μια πολύ σημαντική ε, ε, σημαντικό ρόλο η, κυβέρνηση του σημερινού στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και της ΦΑΡΚ θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει την ερευνευτική αυτή προσπάθεια. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις ε, απόψεις σας για την εξέλιξη αυτή, για τις εξελίξεις στον τομέα της ερευνευτικής ε, διαδικασίας στην Κολομβία και πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Βαλένσια, θα δώσω το λόγο στον κύριο Χορέγγι, για κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία και το μόνο που έχω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, που ήταν πολύ σωστά, δύο πράγματα, λοιπόν, που είναι σωστό να μπουν στην εισαγωγή αυτής της ανταλλαγής απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισημερινού. Ο Ισημερινός είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή, το είπε και ο κύριος Μακάλιστερ, όταν μίλησε για τις δύο χώρες ε, που, με τις οποίες συνορεύεται, Κολομβία και Βενεζουέλα, αλλά είναι σημαντικό ο υπουργό να μας εξηγήσει την πολιτική αλλαγή που λαμβάνει η χώρα στην χώρα του και τι προσανατολισμό έχει ο Λενίν Μορένο, ο πρόεδρος, ε, για, για το εσωτερικό της χώρας και για την κατάσταση στην ε, περιοχή. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ ε, και από μέρους μου και με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ο υπουργό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ για τα πολύ συμπαθητικά σας λόγια και σας κύριε ε, Χαουράκη. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ήρθαμε εδώ πέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις για την ανάπτυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισημερινού. Νομίζω ότι η επευκαιρία, όπως είπε, είπαν και οι δύο προλαλήσαντε, μπορούμε να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τη Λατινική Αμερική και βεβαίω το, η χώρα μου, ο Ισημερινό και βρίσκεται στην περιοχή αυτή, αλλά έχει και ιστορικό ρόλο να παίξει και έχει παίξει στην, ε, στις σχέσεις ε, στην περιοχή. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας με την ε, Ευρώπη. Αν μπορείτε να πλησιάσετε το, στο μικρόφωνο παρακαλώ για να σας ακούμε. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προσέγγιση με την Ευρώπη για λόγω του ότι έχουμε ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς. Έχουμε επίσης από την άλλη κοινά συμφέροντα και στόχους σε διμερές επίπεδο αλλά και σε πολυμερές επίπεδο φυσικά. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σταθώ στη σημασία που δίνουμε στο διάλογο των δύο περιφερειών που πρέπει να αναπτυχθεί μέσω από τον, τις επαφές ΣΥΛΑΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε ένα χώρο για ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε σημαντικέ προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ολοκλήρωση του θεματολογίου 2030 και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόβλημα των ναρκωτικών, η, ανάπτυξη, η στήριξη της ανάπτυξης, πολιτική υπέρ των δύο φύλων και άλλα θέματα γενικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει σημασία αυτό που πιστεύει το ΚΟΕΔΟΡ για τον διάλογο στα πλαίσια της Eurolat, η EULAT επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ομολόγων της Λατινικής Αμερινής, ούτως ώστε να καταλάβουμε αμοιβαία καλύτερα την πραγματικότητά μας και να βρούμε τις συνέργειες για να αναπτύξουμε ε, ένα, ένα θεματολόγιο θετικό που να ενδιαφέρει και τις δύο περιφέρειες αυτές του κόσμου. Από τη στιγμή που ο Λενίν Μορένο ανέλαβε το Μάιο του 2017 την Προεδρία του Ισημερινού, η, η συνεργασία και ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προοδευτικά εντατικοποιήθηκαν. Εγώ ως υπουργό Εξωτερικών του Ισημερινού προωθώ αυτούς τους προσανατολισμούς που επιθυμεί ο κύριος Μορένο προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαν το νέο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα που υπάρχει στον Ισημερινό από τη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Μορένο. Αναφέρθηκε ο κύριος Χαουρέγγι για αυτό το θέμα. Ε, υπάρχει μια εθνική αποδοχή των δεσμεύσεων του Ισμερινού να προωθήσει το διάλογο και να αφήσει στην πάντα την, την τακτική της αντιπαράθεσης για να λυθούν ε, κοινωνικές εντάσεις. Όχι με την επιβολή, αλλά με την δημοκρατική ανοχή και να προωθήσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά σε εκείνες τις κρίσιμες περιοχές όπου στο παρελθόν ε, είχαμε ε, καταπίεση της ελευθερίας έκφρασης, των ατομικών ελευθεριών και της ελευθεροτυπίας. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική συνένεση ε, και αυτό φαίνεται στις σχέσεις μας με άλλες χώρες. Παραδείγματο χάρη, ο ειδικό ε, εισηγητή του ΟΗΕ μας επισκέφθηκε πρόσφατα ε, και μίλησε για την ελευθερία έκφρασης και την επικοινωνία και έδειξε την ε, ατμόσφαιρα σεβασμού αυτών των ελευθεριών που υπάρχει τώρα στο νησιμερινό. Σε κοινωνικό πλαίσιο, η κυβέρνηση του Προέδρου Μορένο επιβεβαίωσε με τις πράξεις, με τη στάση του, το, τη δέσμευση που έχει αναλάβει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία όλων των πολιτών μας και κυρίως εκείνων των ατόμων που είναι πιο ευάλωτα στην κοινωνία μας. Το σχέδιο ανάπτυξης ε, λαμβάνουμε υπόψη τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης και τους στόχους ε, βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Ε, δεδομένων ε, δυσκολιών που έχουμε με τον προϋπολογισμό, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ε, και λόγω των στάσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων ε, και του πώς ε, χρησιμοποίησαμε τα έσοδα από το, τους και το πετρέλαιο που είναι βασικό εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας. Αυτό είναι σημαντικό προϊόν για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις, ε, στις σχέσεις με τον Ισημερινό. Είναι παρούσα η Ευρώπη, ειδικά όταν ήρθαν ε, μαζικά ε, Βενεζουελιάνοι από τη γειτονική χώρα και από άλλες χώρες στη χώρα μας. Τρία εκατομμύρια Βενεζουελιάνοι έφυγαν από τη χώρα τους λόγω της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που υπάρχει. 240.000 ε, Βενεζουελιάνοι ήρθαν στη χώρα μου και έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε την, ε, το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ε, έχουν 100.000 ε, άτομα, έχουν πάρει εργατική στέγη. Ε, επίσης, τους δίνουμε έγγραφα για να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση διαμονής τους στον Ισημερινό και πολιτικές προστασίας της υγείας, ε, τις εργασιακές την ασφάλεια, τα την εκπαίδευση, αυτά με αποφάσεις και ένα πνεύμα πραγματικής αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Στα πλαίσια της ε, περιφέρεια, σε όλη την, ε, με δεδομένη την πραγματικότητα που υπάρχει στην ε, περιφέρεια αυτού του κόσμου, λόγω της κρίσης των προσφύγων από την Βενεζουέλα, ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, το μεγαλύτερο μεταναστευτικό φαινόμενο που έζησε η Λατινική Αμερική ε, στην ιστορία της, δηλαδή εντός της Λατινικής Αμερικής μετακινήσεις πληθυσμών. Μία ομάδα ευρωβουλευτών θα πάνε στο Περού για να διαπιστώσουν την κατάσταση της, των μεταναστών από, το, από τη Βενεζουέλα στην περιοχή. Εμείς στην, στον σημερινό σας προσκαλούμε, ούτως ώστε αυτή η αντιπροσωπεία να μας επισκεφθεί με αντίστοιχο στόχο για να επιστρέψω την κατάσταση στη χώρα μου. Αυτό θα βοηθήσει ούτω ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν μια συνολική θεώρηση για τι προκλήσει που έχουμε λόγω τη μετανάστευση από τη Βενεζουέλα για όλη τη Λατινική Αμερική αλλά και για τη χώρα μου ιδιαίτερω. Και να δείτε τι τεράστιε προσπάθειε που έχει κάνει ο σημερινό για να δείξει αλληλεγγύη με του Βενεζουελιάνους με δημόσιε πολιτικέ απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, στον οικονομικό τομέα έχουμε σημαντικές ε, προκλήσεις ε, να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Ε, η πέμπτη συνεδρίαση της Εμπορικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας Ισμερινού και Περού θα γίνει στον Ισμερινό. Έγινε μάλλον τον Δεκέμβριο του 2018 πριν από λίγες εβδομάδες. Ε, ένα από τα βασικά θέματα ήταν να δούμε, ε, να δημιουργήσουμε την Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και αξιολόγηση των εμπορικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ενισχύσει περισσότερο τις ε, σχέσεις ανάμεσα στις λατινοαμερικανικές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο για την ε, πολυμερή συμφωνία με βάση μια έκθεση της ε, Επιτροπής Εμπορίου τη Ένωση. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια από τη συμμετοχή του Ισμερινού οι εισαγωγές από τη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 10,8% ενώ οι εξαγωγές ε, από την Ευρώπη στον Ισμερινό αυξήθηκαν κατά 36%. Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι ευνοϊκό για το Ισημερινό. Είχαμε 35 εκατομμύρια και, ε, τον, και 156 τον Αύγουστο. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισημερινού και ο διάλογος είναι σημαντικό εργαλείο για αυτό το μέσο για να ξεπεράσουμε διάφορα φράγματα που έχουμε. σε άλλου τομεί των οικονομικών σχέσεων Ισημερινού ε, και Ευρώπης ε, βλέπουμε με αισιοδοξία τις συζητήσεις που έγιναν, ξεκίνησαν το Μάιο ε, στην περιοχή, ούτω ώστε να προωθήσουμε ε, με τις διμερείς συμφωνίες τις επενδύσεις ε, προς όλες τις χώρες. Παρότι το θέμα είναι διμερούς χαρακτήρα, τις σχέσεις δηλαδή, του Ισημερινού με διάφορες χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οι συμφωνίε πρόθεση των επενδύσεων μπορούν να οριστικοποιηθούν σε, στο εγγύ μέλλον και θα συμπληρώσουν τι πολιτικέ ε, ανάπτυξη και επενδύσεων του Προέδρου Μορένου. Ε, θα βοηθήσουν τι επενδύσει ε, μέσω και φορολογικών διευκολύνσεων και θα ενισχύσουν την νομισματική σταθερότητα της χώσης και θα μας φέρουν εξωτερικές επενδύσεις που θα φέρουν πρόοδο, οικονομική ευημερία, απασχόληση στη χώρα μου. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, επ' ευκαιρία θα ήθελα να πω ενώπιό σας ότι παρότι το θέμα συζητείται σε, άλλους, σε άλλα φόρουμ της ε, ε, Ένωσης γενικά, ε, εμείς ελπίζουμε να μας δοθεί εξαίρεση από την υποχρέωση των θεωρήσεων σε περίπτωση που οι θεωρήσει αυτής είναι βραχίας διάρκειας. Είναι πολύ σημαντική ε, η στάση του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, υποστηρίζουν πολλές χώρες, ε, πολλές κυβερνήσεις δηλαδή, την διευκόλυνση αυτή προς τον Ισημερινό, γιατί έχουμε πολλούς δεσμούς. Πολιστικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ. Επίσης, εμείς δεν θα ζητάμε θεωρήσει από τους Ευρωπαίους πολίτες που μας επισκέφτονται για σύντομη διάρκεια. Εξαιρετικές είναι οι σχέσεις μας και έχουμε και πολυμερές εμπόριο. Ε, α, όλα αυτά θα βοηθήσουν τις ανταλλαγές Ευρώπης και Ισημερινού και θα διευκολυνθεί και από την εμπορική συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την στήριξη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, για το θέμα αυτό. Ε, χαιρετίζω όλους, κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Your Excellency, thank you for your... Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε για την ε, αρχική σας τοποθέτηση, για το τι σημαίνει στη χώρα σας και στην ε, Νότιο Αμερική. Και τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο για μια ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, συνάδελφοι, αν θέλετε τον λόγο, κάντε μου ένα νόημα. Ο κύριος Αλαφράγκα, λοιπόν, έχει πρώτος τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για τις σημαντικές πολιτικές αλλαγές που έχετε καταφέρει και επίσης για τις δράσεις αλληλεγγύης που έχει λάβει η χώρα σας σε αυτή τη σύγκρουση έναντι των προσφύγων. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να αναγνωρίσω τις πολύ σημαντικές προόδους που έχει επιτύχει ε, η χώρα σας και τα αποτελέσματα που έχουμε διαπιστώσει στον τομέα του εμπορίου. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ε, και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και αντίστοιχη βελτίωση των επενδύσεων. Αυτό είναι απολύτω απαραίτητο. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, μια και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την θέση σας για το ζήτημα της Βενεζουέλας και σε σχέση με την αναγνώριση του μεταβατικού πρόεδρου. Θα ήθελα επίσης να με ενημερώσετε για διάφορες αναφορές για ξενοφοβικές πράξεις ή πράξεις ε, αντικδίκησης που διαπιστώθηκε ότι συνέβησαν σε ορισμένες γειτονικές χώρες. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε πώς βλέπετε το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής, δεδομένων των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην ε, περιοχή σα και δεδομένων επίση επίσης των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Από του σοσιαλιστέ, η κυρία Άννα Σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρέμβασή σας στην Επιτροπή μας. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να εμβαθυνθούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η σημερινού προς όφελος της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης από κοινού των διαφόρων προκλήσεων που έχουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Έχει διάφορες επιπτώσεις ε, οι οποίες επηρεάζουν όλες τις ε, χώρες της περιοχής. Αυτή η εσωτερική κρίση στη Βενεζουέλα έχει επηρεάσει όλες τις όμορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και ο σημερινός. Μιας και πολλοί πρόσφυγες καταφεύγουν στη χώρα σας. Αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε ότι πρόκειται να γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην περιοχή, αλλά και επίσης σε διεθνές επίπεδο. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η θέση της ε, διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο πρόεδρος Μαδούρο να οργανώσει εκλογές οι οποίες να πληρούν τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και ε, νομιμότητας. Ε, είναι αυτό εξάλλου ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. ρωτώ, είναι επίσης, θα χρειαστούν επίσης διεθνείς παρατηρητές. Ρωτώ. Επίσης θα ήθελα να εισφέρω και ακόμα μία διάσταση στη συζήτηση αυτή που έχει σχέση ε, με την υποστήριξη που δείχνει η Ρωσία στην κυβέρνηση Μαδούρο συμπεριλαμβανομένης και της στάθμευσης ε, σε ε, έδαφος της Βενεζουέλας πυρηνικών βομβαρδιστικών το θέμα αυτό το έθεσε και ο συνάδελφος Σαλαφράγκα, το, έχουμε, το έθεσα και εγώ ε, και ε, έχει σχέση με την κατάσταση στην Ικαράγουα. Μια χώρα γειτονική με τη δική σας, η οποία και εκείνη έχει υποστεί τα δεινά της καταπίεσης. Και εδώ ούτε οι χώρες της περιοχής, ούτε η διεθνής κοινότητα διαπιστώνω να έχει κινητοποιηθεί για να υποστηρίξει το λαό της Νικαράγουας και να ζητήσει διάλογο, να ζητήσει εκλογές, έτσι ώστε να διοργανωθούν εκλογές. Ελεύθερες, ε, με διαφάνεια και με διεθνείς παρατηρητές. Τα γεγονότα στην Νικαράγουα ήταν δραματικά, ήδη από τον Απρίλιο. Ε, έχουμε επισκεφθεί πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές. Είχαμε τη δυνατότητα πράγματι, όμως συνεχίζεται η καταπίεση και είναι πολύ, πολύ ουσιαστική, πολύ, πολύ δραματική. Πώς γίνεται λοιπόν οι χώρες της περιοχής να μην έχουν κινητοποιηθεί για μια αντίστοιχη λοιπόν κατάσταση. Και εδώ είχαμε απέλαση των εκπροσώπων του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, του εκπροσώπου του, του, του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Γνωρίζουμε τις ε, σημαντικές ε, εξελίξεις και την σημαντική βελτίωση που έχει σημειωθεί στη χώρα σας. Μας τα περιγράψατε συνοπτικά. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπορική συμφωνία, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Ισημερινός, όπως και η Κολομβία, θα μπορέσει να ε, συνεργαστεί καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που ακούω ότι και τα αριθμητικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Και αυτό μπορεί να ενισχύσει και τον πολιτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι επίσης που έχετε προσπαθήσει να εντάξετε στις πολιτικές σας ε, τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030 και να δώσετε έμφαση στις κοινωνικές πολιτικές. Και σε, αυτόν το, σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρασταθεί στο πλευρό σας. Οι συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν ε, στο θέμα της Βενεζουέλας και της ε, Νικαράγουα ιδιαίτερα σε σχέση με τη Βενεζουέλα. Αναφέρθηκε η επιρροή της Ρωσίας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τι πιστεύετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Κίνας αυτή τη στιγμή. Και επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Πιστεύετε ότι με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες η Κίνα θα μπορούσε να ασκήσει μια κάποια επιρροή ώστε να υπάρξουν αλλαγές στην Πενεζουέλα. Τι εννοώ. Το γεγονός ότι η Κίνα έχει εμπορικέ σχέσει με άλλε χώρε τη Λατινική Αμερική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε η Κίνα να αλλάξει τη θέση τη σε σχέση με τη Βενεζουέλα, δεδομένου ότι και η Ρωσία και η Κίνα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στι εξελίξει στο, στο, στο, θέμα αυτό, στην κατάσταση στη χώρα αυτή. Επίση, Ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο μελλοντικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερθήκατε στο ζήτημα των θεωρήσεων σίγουρα, και επίσης πώς εκρίνεται τον μηχανισμό παρακολούθησης της εμπορικής συμφωνίας ε, η σημερινού Ευρωπαϊκή Ένωση. θεωρείται ότι λειτουργεί, μπορούμε να τον βελτιώσουμε και επίση. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσει στον Ισημερινό γνωρίζουν τι ευκαιρίε που του δημιουργεί που τους δίνονται με αυτή την συμφωνία. Και τέλος θα ήθελα για άλλη μια φορά να σα συγχαρώ για την ανθρώπινη και εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσετε στους πρόσφυγες που έρχονται από τη Βενεζουέλα στη χώρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπιλμπάου. Τελευταίος ομιλητής, κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και σας ε, κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε για, σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Εξωτερικών και με την αντιπροσωπεία εδώ, των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την Συμφωνία Σύνδεσης ε, για τον σημερινό Περού και Κολομβία. Θεωρώ ότι ήταν το αποτέλεσμα μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία διαπραγματεύσεων ε, και την ε, αυτόνομη κίνηση του σημερινού που ξεκίνησε να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση αϊφόρου κατεύθυνση και βέβαιω με την Συμφωνία Σύνδεσης συμφωνήθηκαν κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα δημερώς που ακριβώς ε, δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει η προσέγγιση αυτή του σημερινού και στο μέλλον και είναι σημαντικό στο μέλλον ε, και να υπάρχει αυτή η πολυμερής ε, προσέγγιση των εμπορικών σχέσεων. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Βολιβία δεν ε, συμμετέχει σε αυτήν την περιφερειακή συμφωνία εμπορίου, αλλά βεβαίως ε, οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει πάντα να εξυπηρετούν την ανάπτυξη της οικονομίας, τους ανθρώπους, ε, την διαφοροποίηση των εθνικών οικονομιών και θεωρώ ότι ο σημερινός εδώ πέρα έχει να επιδείξει ακριβώς μια επιτυχή τέτοια διαφοροποίηση της ε, οικονομίας. Ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξάρτησης ε, από το πετρέλαιο που δεν είχε ξεπεραστεί εδώ και δεκαετίες και είναι και μία από τις αιτίε για την περίπλοκη κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς βλέπετε τις ε, δυνατότητες αυτές στην Λατινοαμερικανική Ήπειρο. Έχουμε και την ε, Βραζιλία. Είδαμε και τι έγινε με αυτό το φρικτό ατύχημα. Ε, Ακριβώ το να μπορέσουμε να φύγουμε, να υπάρξει μια πυκλομορφία, να διαφυλαχτούν και οι θέσει εργασία και το περιβάλλον. Ο πρόεδρο ο Βολσονάρο ανακοίνωσε πως θα αρχίσει η υλοτομία, υπεραιτέρω υλοτομία στον Αμαζόνιο και η Γεωργία. Αυτό όμως σημαίνει ότι κινδυνεύει ένας από τους πράσινους ε, πνεύμονες του πλανήτη, δηλαδή έχει παγκόσμια σημασία και έχει σημασία άρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα αναπτύξει την παγκόσμια εμπορική πολιτική της για να υπάρξει μια διαφοροποίηση και πώ θα μπορέσουμε και εμείς να την βοηθήσουμε. Δηλαδή, γιατί αφορά άμεσα το μέλλον μας. Ναι, δηλαδή, είχαν ξεκινήσει κάποια έργα με τη Sony και την ITT ε, στον Ισημερινό, τα οποία δεν είχαν προχωρήσει καθόλου. Λοιπόν, και επιτρέψατε μου να σας πω πως ε, εμείς ε, στην ομάδα μας ε, σας υποστηρίζουμε να υπάρξει ακριβώ το θέμα αυτό το οποίο θέλετε με την βίζα για την ζώνη Σέγγεν και δεν θέλουμε να υπάρχουν εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής ε, απέτηση που απευθύνουμε προς το Συμβούλιο, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Περού και Κολομβία το έχουν αυτό, την, την βίζα. Γιατί να μην έχει και ο Ισημερινός. Και τέλος ναι, βεβαίως είμαστε αλληλέγγυοι μαζί σας γιατί εδώ και δεκαετίες φιλοξενείτε πρόσφυγες από την Κολομβία. Η ειρηνευτική διαδικασία εκεί πέρα δεν έχει τελειώσει. Αυτό σημαίνει πως αυτό το οποίο γίνεται και με τους πρόσφυγες από την Βενεζουέλα ακριβώς μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία, γιατί δεν ξέρουμε βεβαίω και αν ο νέο Κολομπιανό πρόεδρο αποτελεί εγγύηση για την ειρηνευτική διαδικασία και θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με την υποκατάσταση τη καλλιέργεια κόκα με κάποιο άλλο προϊόν και βέβαια έχουμε όλε αυτέ τι μεθοριακέ περιοχές ε, ε, ε, και η σημερινού και το τι μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα για να αντιμετωπίσετε αυτά τα φαινόμενα και το τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε όσον αφορά τα γεωργικά σας ε, προϊόντα. Γιατί βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τη δική σας σταθερότητα και την ασφαλεία σας ε, στην χώρα και θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο άλλο τώρα που ζήτησε τον λόγο. Δίνω τον λόγο και πάλι στην κυρία Μαριάν Φανστέιν, η οποία είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στον Ισημερινό. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι κύριε Υπουργέ που βρίσκομαι εδώ και σας έχουμε στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα κάνω ερωτήσεις, δεν θα απαντήσω εγώ σε ερωτήσεις. Ε, θα το κάνετε εσείς φαντάζομαι σε λίγο. Θα ήθελα απλά να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών στο εξή. Ε, είμαι εδώ και δυόμιση χρόνια τώρα στον Ισημερινό. Ο Ισημερινός έχει αλλάξει. Δεν θα αναφέρω όλες τις αλλαγές που έχω δει γιατί είναι πάρα πολλές. Θα ήθελα απλά να επισημάνω το εξής, μία αλλαγή που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική. Ο διάλογος, η ελευθερία έκφρασης, πράγματα καινούργια στην χώρα. Όταν έφτασα εγώ είχα την αίσθηση ο κόσμος φοβόταν να μιλήσει. Φοβόταν τις κυρώσεις, ε, υπήρχε ένας νόμος ε, περί επικοινωνίας που ήταν πάρα πολύ δύσκολος ε, και έκανε δύσκολη τη δουλειά των ΜΜΕ Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Βεβαίως ε, αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τους Ευρωπαίους γιατί για μας ε, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αυτό η ελευθερία έκφρασης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το νέο πνεύμα άλλαξε ολόκληρη την ε, εικόνα της χώρας και φαίνεται αυτό και στις διεθνείς σχέσεις και πάλι δεν θα επεκταθώ σε σχέσει με τις γειτονικές χώρες ή με την Κίνα ή τη ΣΥΠΑ. Απλά να πω το εξής. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας έχουν προχωρήσει πολύ τους τελευταίους 18 μήνες που κυβερνά ο πρόεδρος ε, Μορένο. Εάν δούμε την εμπορική συμφωνία, μια τεράστια επιτυχία, δεν το περιμέναμε ποτέ ότι μόλις μετά από ένα χρόνο θα βλέπαμε αύξηση κατά 20% των εμπορικών ροών. Εντάξει, ο δεύτερο έτος ήταν κάπως μικρότερη, αλλά προχωράμε προς την εφαρμογή αυτή της συμφωνίας και την εκμετάλλευση όλων των ε, ευκαιριών που προσφέρει στη χώρα. Δεύτερον, η συνεργασία. Πριν από δύο χρόνια υπήρχε πολύ μικρή ικανότητα απορρόφησης το διμερές πρόγραμμα που έχουμε μπορεί να επεκταθεί και μέχρι το 2020 και πέρσι είχαμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε πολύ στενά με την κυβέρνηση του σημερινού και ειδικά το Υπουργείο Εξωτερικών και πριν από δύο μήνες είχαμε την συμφωνία των 28 κρατών μελών για 25% του διμερούς φακέλου. Θα μπορέσουμε λοιπόν έτσι να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν για να επανενεργοποιηθούν οι περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό του 2016 εφενός. Από την άλλη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στα βόρεια σύνορά της. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά και καταλήγω λέγοντας ότι και στο πολυμερές επίπεδο έχουμε δει ένα σταδιακό άνοιγμα όσον αφορά την ευθυγράμμιση της θέσης ε, του Ισημερινού, ειδικά με εμάς, ε, οπωσδήποτε, ε, και σε άλλα φόρα. Και είναι πάρα πολύ θετικό το να βλέπουμε πως μόλις σε 18 μήνες μπορέσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας σε όλα αυτά τα θέματα. Και πρέπει να το ξέρουν αυτό οι ευρωβουλευτές. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων για το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για την βελτίωση των σχέσεων των χωρών μας το τελευταίο 1,5 έτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φανστέιν. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε διάφορες ερωτήσεις. Τέλος, να προσθέσω και εγώ δύο ερωτησούλες. Οφορούν δύο χώρες που δεν είναι ε, άμεση γειτονές σας, δεν συμμαρεύεται. Η μία είναι η Βραζιλία. Μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε τη νέα πολιτική κατάσταση στη χώρα και ειδικά ως κάποιος ο οποίος γνωρίζει τη βραζιλιάνικη νοοτροπία και της νέας κυβέρνησης πώς θα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να συνεργαστούμε με τον νέο Βραζιλιανό πρόεδρο. Και δεύτερον, ε, η χώρα σας αναγνώρισε τον κύριο Κουάντο ε, μεταβατικό. μεταβατικό πρόεδρο. Τι προτείνεται σε εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το πολύ λεπτό θέμα. Eh, Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές και σας κύριε Μακάλιστε για τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Θα ήθελα να τις ομαδοποιήσω τις απαντήσεις για να με φτάσει και ο χρόνος. Θα ξεκινήσω από τις ερωτήσεις του κυρίου Ιγνάσιο Σαλαφράγκα ο Ισμερινός αναγνώρισε τον ε, ενδιάμεσο, το μεταβατικό πρόοδο, τον κύριο Γκούια εδώ. Και το κάναμε λόγω του τι συνέβη την, το Μάιο του 2018 στην εκλογική διαδικασία. Ε, διαδικασία που οδήγησε στην ανανέωση της του Μαδουρού. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και παρατυπίες, ε, όπως είπαν οι διεθνείς παρατηρητές της ε, εκλογές της ε, Βενεζουέλας. Σοβαρά προβλήματα, σοβαρές αντιρρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε στην οργάνωση των Αμερικανικών κρατών να θεωρήσουν ότι θα πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα, ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε ή να μην αναγνωρίσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή ήταν μια πρώτη ιδέα που ακούστηκε και τελικά ε, δείχνει πόσο δεσμευμένοι είμαστε απέναντι στην δημοκρατία στην ε, Βενεζουέλα και στην, στην προσπάθεια επίλυσης των κρίσεων που υπάρχουν ε, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο στη χώρα. θέσαμε αυτό το ερώτημα, αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για αυτά τα θέματα των εκλογών. Συνεχίσαμε όμως με αυτή την στάση, με αυτή την άποψη. Και στις 10 Ιανουαρίου, όταν ο Μαδούρο ανέλαβε ξανά την Προεδρία, αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε στην τελετή. Μία εβδομάδα ή λίγες μέρες πριν, είμαστε παρόντες στη συνέλευση των, Αμερικανών, των Αμερικανικών κρατών ε, για το θέμα αυτό της ε, διαφάνειας ε, στην Βενεζουέλα. Ε, εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να αναμειγνιόμαστε σε εσωτερικές υποθέσεις. Θεωρούμε ότι οι διεθνείς δράσεις για να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ισοδυναμεί με παραβίαση της βασικής αρχής αυτής του διεθνούς δικαίου, της μη παρέμβασης δηλαδή σε τορικές υποθέσεις ενός κράτους. Εξάλλου, εμείς συμφωνούμε με το χάρτη ιδεοντολογίας που υπογράφηκε το 1980 μεταξύ διαφόρων χωρών της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων και η Βενεζουέλα, μια δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, για λόγους τέτοιου, για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θεωρούμε ότι αυτή η παρέμβαση ισοδυναμεί με παρέμβαση τι εσωτερικής υποθέσεις ενός κράτους. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που μεταξύ άλλων που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε ε, δεσμευτεί να το σεβαστούμε αυτό το εργαλείο και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη. Εν συνεχεία, υπάρχουν ανησυχίε που εκφράστηκαν από ευρωβουλευτέ γιατί σε διάφορε χώρε τη Λατινική Αμερική ε, υπάρχουν ε, ξενοφοβικές τάσεις απέναντι στους ε, μετανάστες από τη Βενεζουέλα και στην βενεζουελιάνικη διασπορά. Αυτές οι ξενοφοβικές τάσεις είναι απομονωμένες. Ο γενικός κανόνας είναι υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών. Τους δίνουμε τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να εγκατασταθούν στις χώρες υποδοχής. Παρά τις τεράστιες ε, οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες που έχει τουλάχιστον ο Ισημερινός, εμείς ε, στεναρά είπαμε ότι οποιαδήποτε δράση κατά των βασικών δικαιωμάτων των ε, ανθρώπων η ηθαγένεια θα καταδικαστούν, θα τις δεχτούμε, θα τις καταδικάσουμε και, και τέτοιες συμπεριφορές και αντίστοιχες συμπεριφορές λοιπόν τις καταδικάζουμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε ούτως ώστε οι μετανάστες αυτοί να έχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις Έχουμε υποδεχθεί χιλιάδες παιδιά από την Βενεζουέλα στα σχολεία μας, έχουν εμβολιαστεί διάφορα παιδιά και 100.000 έχουν μόνιμη ε, θεώρηση ε, για να ζήσουν μόνιμα στο Ισημερινό. 40% του συνολικού πληθυσμού των προσφύγων ε, από τη Βενεζουέλα έχουν πάρει αυτά τα χαρτιά και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία τακτοποίησης ε, της κατάστασής τους γιατί έχουμε αναλάβει αυτή την ε, ανθρωπιστική δέσμευση απέναντί τους. συνεχεία, κυρία Ναγκόμες, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Ποιο είναι το μέλλον, τι μας περιμένει. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δίνουμε μεγάλη έμφαση στον Ισημερινό, στο να υπάρχει, στο να δοθεί λύση δημοκρατική στη Βενεζουέλα, η οποία δεν θα αποκλεί κανέναν από τους βασικούς φορείς εντός και εκτός της Βενεζουέλας στη διαδικασία αυτή. Χωρίς αποκλεισμούς λοιπόν λύση, μία λύση η οποία θα γίνει μέσα σε ατμόσφαιρα αποκλεισμό δεν υπάρχει αυτό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αδύνατον να προχωρήσει μια εκλογική διαφανής διαδικασία. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν διαφανείς εκλογές με σεβασμό του κράτους δικαίου. Ε, πιστεύουμε στη σημασία των διεθνών παρατηρητών για να δοθούν οι απαραίτητες ε, εγγύησεις. Αυτές είναι οι βάσεις για να γίνει η δημοκρατική αναδιάρθρωση της χώρας. Συμφωνούμε με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούμε αυτή τη δημοκρατική λύση μέσα από ελεύθερες εκλογές. Πιστεύουμε ότι η μοναδική λύση και ο πρόεδρος, ο δικός ο Γουαϊδό ε, ακριβώς αυτό θέλει, ούτω ώστε να φτάσει σε σταθεροποίηση η χώρα και να επανέλθει σε μια κανονική θέση, να τακτοποιηθεί το οικονομική της κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ρωσία η παρουσία της Κίνας εκεί. Είναι μία από τις άλλες ερωτήσεις που ακούσαμε από την κυρία Μπιλμπάου. Εμείς πιστεύουμε ότι η δράση από άλλες χώρες της διεθνούς κοινότητας ε, απέναντι στη Βενεζουέλα μπορούμε να είναι θετικές, αλλά όχι από μόνες τους. Αλλιώ δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορούν οι άλλοι να λύσουν το πρόβλημα για τη Βενεζουέλα. Ο, το κράτος της Βενεζουέλας, ε, η αντιπολίτευση ε, και όλοι οι φορείς μπορούν να φτάνουν σε μια συνεννόηση. Τώρα, καμία στάση από εξωτερικούς φορείς δεν μπορεί να βρει τη λύση. Πιστεύουμε σε μια, οικονομική, σε μια επικοδομητική δράση της διεθνούς κοινότητας, στηρίζοντας τον εθνικό διάλογο στη Βενεζουέλα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας διεθνής διευκολυντής για τη Λατινική Αμερική, ε, στο διάλογο δηλαδή, ήταν πολύ επωφελής ε, στο παρελθόν σε κρίσιμες περιπτώσεις σε χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής, τη δεκαετία του 80 και 90. Ας πούμε η δράση της ομάδας του Ρίο για να υπάρξει συμφωνία στην Ικαράγουα, Γουατεμάλα και Αλσαλβαδόρ. Γιατί όχι και στη Βενεζουέλα. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, μια ομάδα επαφής ε, των χωρών αυτών ε, για και οποιαδήποτε στιγμή δημιουργηθεί θα στηρίξει το, η χώρα μου, η αυτή την ομάδα ούτως ώστε αυτή η ομάδα εθνών ε, της διεθνούς κοινότητας να προωθήσει τα απαραίτητα μέτρα. Νικαράγουα. Είναι μια ανησυχία που και για μας Ήμασταν πολύ δραστήριοι από τις πρώτες ε, διαδηλώσεις που καταπνίγηκαν ε, από τον πρόεδρο Ορτέγα, 400 ε, νεκροί, χιλιάδες κρατούμενοι στις διαδηλώσεις αυτές, υπερβολική χρήση βίας που, κατα... που καταρρύπτει διάφορες αρχές των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι ο εθνικός διάλογος στην Καραγουά είναι η μόνη λύση, μια δημοκρατική λύση. Ξανά, υπάρχει μια, ένας παραλληλισμός, ας πούμε, τη Βενεζουέλα. Νικαράγουα, Βενεζουέλα. Βλέπουμε κάποιες παράλληλες πορείες. Πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση και θα πρέπει τελικά και στην Νικαράγουα να εκφραστούν οι πολίτες ούτω ώστε να ε, αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη στη χώρα και να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με τις χώρες ε, της περιοχής, γιατί είμαστε μέλο της ομάδας εργασίας του Μονίμου Συμβουλία της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών για την Ικαράγουα και με μεγάλη ανησυχία είδαμε και καταδικάσαμε την κατάσταση και είπαμε μέσα από την οργάνωση Αμερικανικών κρατών ότι δεν είναι αυτή η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα πρέπει η λογική, ε, η δημοκρατική, ο δημοκρατικός διάλογος να πρετανεύσει. Σχέση με αυτά που ρωτούσε η κυρία Πιλπάου, Μιλήσαμε ήδη για την Ικαράγουα και μιλήσαμε ήδη για τα επιρροή που μπορεί να έχουν άλλα κράτη. Με ρωτήσατε όμως επίσης ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και των άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Πιστεύουμε ότι όλε αυτέ τι χώρε τη Λατινική Αμερική μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε τελικά να βρεθεί μια δημοκρατική λύση στο πρόβλημα τη Βενεζουέλα. Και υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο, σε αυτή τη συζήτηση. Ο σημερινό θεωρεί ότι μια σύγκρουση τόσο περίπλοκη όσο αυτή της Βενεζουέλας είναι μια σύγκρουση η οποία δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με έναν διάλογο ουσιαστικό, με στόχους, έτσι ώστε να βρεθεί μια δημοκρατική λύση. Μόνο έτσι. Το να κάνουμε ένα διάλογο χωρί να αναζητούμε δημοκρατική λύση θα ήταν απλώ χάσιμο χρόνο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει καλή θέληση από όλε τι πλευρέ και να υπάρχει η διάθεση να βρεθεί μια λύση στην οποία να μπορέσουν να συμφωνήσουν όλοι οι Βενεζολάνοι. Πιστεύω ότι αν βρεθεί μια τέτοια λύση θα τύχει τη υποστήριξη των περισσότερων κρατών της Λατινικής Αμερικής. Πολλά κράτη της περιοχής έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αναγνωρίζοντα το μεταβατικό πρόεδρο εδώ, τονίζοντα όμω ταυτόχρονα ότι η υποχρέωση του θα είναι στο, όσο δυνατόν γρηγορότερα να οργανώσει πραγματικά συμμετοχικές ε, έντιμες ε, και εκλογές με διαφάνεια. Αυτή είναι μια θέση πιστεύω έχει εκφραστεί ουσιαστικά στην περιοχή. περάσουμε τώρα από το ζήτημα της Βενεζουέλας και της Κολομβίας και γενικώ τα ζητήματα τα περιφερειακά τη γενικότερη συζήτηση περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όπως ανέφερε και η κυρία Πρέσβης, έχουμε μια θετική αξιολόγηση της λειτουργίας της συμφωνίας. Η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τη θεωρούμε μονάχα μια εμποριακή ε, συμφωνία, το είπε είναι ένα μέρος ε, των πολυσχεδών σχέσεων που θέλουμε να αναπτύξουμε μεταξύ σημερινού και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε να διαμορφωθεί ε, μία ε, σχέση που να συμπεριλαμβάνει πολλά αλληλένδετα μεταξύ του ζητήματα και την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Καθώς επίσης και την προσπάθεια που θα κάνουμε από κοινού να επιτύχουμε κοινού στόχου, όπω για παράδειγμα την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντο, την κοινωνική προστασία κτλ. Έτσι λοιπόν και από αυτό το πρέγισμα θεωρεί ο σημερινό ότι η συμφωνία λειτουργεί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στο χέρι του Ισημερινού, του Περού, της Κολομβίας για να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτός ο πολυμερής μηχανισμός εμπορικών σχέσεων να αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί συνολικά η σχέση των χωρών αυτών αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η συμφωνία, αυτή η σχέση. Όπως έλεγα, δημιουργήθηκε η συμβουλευτική ομάδα στην οποία, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντική και πολύ θετική αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ε, πολυμερή εμπορική συμφωνία, γιατί δίνει μια δημοκρατική δημοποίηση και μια λογοδοσία. Έρχομαι σε ορισμένα από τα ερωτήματα του κύριου Σούλτς. Σύντομα. Βεβαίω, το Εκουαδόρ, το, το Ισοημερινός, επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. Και βεβαίω αναμένουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση από άλλε χώρε όπω η Βολιβία για να δημιουργηθούν τέτοιε πολυμερεί συμφωνίε. Εμείς έχουμε υποστηρίξει τον λαό της Βολιβίας στο παρελθόν και συνεχίζουμε να το πράττουμε, πιστεύουμε ότι αν βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει μια πολυμερή συνεργασία και βεβαίως ε, ε, σεβόμενοι ότι το γεγονό ότι αυτή την απόφαση θα πρέπει να τη λάβει ε, η Εθνικά Κυρίαρχη Βολιβία, εμείς είμαστε ανοιχτοί και το καλωσορίζουμε ως ενδεχόμενο. Τώρα το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζουμε ως είναι το τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο. Γνωρίζετε ότι είναι ευχή και κατάρα η ύπαρξη υδρόγων ανθράκων σε μια περιοχή, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε κάποιους τομείς της οικονομίας. Επιδιώκουμε μέσω των οικονομικών σχεδίων που έχουμε και των αλλαγών που προσπαθούμε να φέρουμε στην διάρθρωση της οικονομίας και της ε, χρήσης του ενεργειακού μείγματος, προσπαθούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Ε, ε, η οποία είναι υπερβολική, δεν, ε, δεν το αμφισβητούμε. Όμως δεν γίνεται μια χώρα όπως η δική μας να έχει να εξαρτάται οικονομικά από κάποια λίγα εξαγωγήμα προϊόντα. Γιατί αυτό δημιουργεί μια σειρά κινδύνους οικονομικούς. Σε εξωτερικές μας οικονομικές μας σχέσεις και αυτούς τους κινδύνους προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε αν θέλετε την οικονομία μας. Και το, η πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μια, ένα εργαλείο γι' αυτό. έτσι ώστε να μεταβούμε από την παλαιότερη σχέση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καινούργια σχέση που είναι αυτή που περιγράφει η Πολυμερή Συμφωνία. Βραζιλία και αποψήλωση των δασών και περιβάλλον. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι, σημαντικός είναι ο Αμαζόνιος. Γνωρίζετε ότι ε, ένα μέρος της Αμαζονίας βρίσκεται στον Ισημερινό. Πόσο μεγάλη είναι η σημασία του για το περιβάλλον. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τη Βραζιλία και όπως έλεγε και ο κ. Μακάλιστερ, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών στην περιοχή του Αμαζονίου. Έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές επαφές, διερευνώντας το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συνθήκη για τη συνεργασία μεταξύ των ημών ε, και των άλλων τεσσάρων κρατών της περιοχής του Αμαζονίου, έτσι ώστε να προστατεύσουμε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη, ευάλωτη και πάρα πολύ σημαντική επίσης για το περιβάλλον, για το, για το περιβάλλον, για τους λαούς μας, για τους ε, αυτόχθονες πληθυσμούς που ζουν στις περιοχές αυτές. Πρέπει λοιπόν εδώ να ε, βρούμε συμβιβαστικέ λύσεις έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική προστασία της περιοχής του Αμαζονίου. Για άλλη μια φορά το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί τίθενται πολλά ζητήματα, πολλές, ε, πολλά διλήμματα, πολλέ αποφάσει που πρέπει να πάρουμε και στι οποίε πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση τη περιοχή ε, για παραγωγικού και οικονομικού σκοπού και στην προστασία του περιβάλλοντο. Ελπίζουμε να βρούμε ουσιαστικέ λύσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχω δύο λεπτά. Μου επιθυμίζει ο πρόεδρο. Γρήγορα, λοιπόν. Σα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, πρέσβη ε, Στέιν για τα καλά τη λόγια και για την υποστήριξη. Έχετε σωστά αντιληφθεί το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει ο σημερινό στη σχέση του με το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με αμοιβαία κατανόηση γιατί αυτό πιστεύω ότι θα ε, βοηθήσει και τους πολίτες του σημερινού και τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προσπαθούμε να χτίσουμε αυτή τη σχέση πάνω σε στερεές βάσεις. Και τέλος, κύριε Μακάλιστερ, τι να σας πω στην ερώτηση που με θέσατε. Είναι δύσκολο να κάνω μια ε, δική μου πρόταση, εκτίμηση για το τι θα πρέπει να γίνει για τον κύριο Γουαϊδό. Ε, πάντως, κατά την άποψή μου, ο σημερινός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής μοιράζονται κάποιες θεμελιώδεις αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, οποιαδήποτε μας προσέγγιση, οποιαδήποτε μας θέση θα πρέπει να την ε, θεμελιώσουμε σε αυτά. Έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς ε, φορείς στην ε, Βενεζουέλα να βρουν τη λύση που χρειάζεται να βρεθούν για τη χώρα τους επί τη βάση των αρχών που όλοι μοιραζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος ε, του συναδέλφου του κύριου Ατόντο που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Νομίζω πως οι ερωτήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη γωνιά του κόσμου για τα όσα συμβαίνουν στην χώρα σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην νέα σας εξωτερική πολιτική. Ε, έχουμε νομίζω κάποια κοινά συμφέροντα και κοινέ θέσει. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και εύχομαι σε εσά και στην πρέσβυρα ε, καλή διαμονή στις ε, Βρυξέλλες και παραγωγική. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρακλήσή σας.